Πρόεδρο, μια και περιμένουμε την εισηγήτρια, την κυρία Γιαννάκου, για την έκθεση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, μου είπαν ότι φτάνει. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την συνάντηση των συντονιστών. Θα σας μιλήσω λοιπόν σχετικά με την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση να μην ε, προχωρήσουμε στην ψηφοφορία το θέμα των άρθρων 49 και 50 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σας το κοινοποιώ λοιπόν αυτό. Και θα σας πω δύο λόγια, μια και περιμένουμε την κυρία Γιαννάκου. Εγώ θύμισα ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί ο πρόεδρος Σούλτς ε, ε, ε, ανέθεσε στην Επιτροπή μας να συζητήσει αυτή την τρομοποίηση η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο σεμιναρίου των Προέδρων τα πρακτικά της οποίας συνεδρίασης σας έχουν υποβληθεί ε, κυρίως σχετικά με το άρθρο 49. Εγώ είχα δεχτεί την έκθεση αυτή και είχα δεχτεί ως ε, συνηθισμένη επιλογή την ε, υποβολή τροπολογιών αντί ε, γνωμοδότησης από την υπεύθυνη για γνωμοδότηση Επιτροπή έτσι ώστε να γίνει πιο απλή η διαδικασία. Μία άλλη δε τροποποίηση είχε προταθεί του άρθρου 50 δηλαδή οι επιτροπές οι οποίες έχουν αναλάβει να εκπονήσουν γνωμοδότηση να μπορούν, λέω, να συμμετέχουν και αυτές οι υπεύθυνες για Επιτροπή σε όλες τις διαδικασίες μέχρι τον τελικό τριμερή διάλογο και την, ε, ε, ε, και την συνδιαλλαγή μαζί με τον πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής πάντα και επίσης να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίες που ε, η αρμόδια επί της ουσίας ε, επιτροπή θα ε, έπρεπε να λάβει υπόψη. Αυτά είχαν καταγραφεί τον Φεβρουάριο της προηγούμενης χρονιάς, αυτή η συνεδρία των Προέδρων στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Και ε, συμπεριλήφθησαν στην έκθεση, την οποία τώρα, όπως σας είπα, δεν θα ψηφίσουμε. Γιατί οι συντονιστές εξέφρασαν την άποψη ότι θα έπρεπε η επόμενη θητεία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την ε, δική μας εμπειρία και τα όσα μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Ο πρόεδρος Σούλτς ε, μας ε, έστειλε δύο επιστολές ε, επιθυμώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε αυτήν τη θητεία. Μάλιστα στην τελευταία επιστολή του έγραφε ότι είναι απολύτως σημαντικό να ολοκληρωθεί σε αυτή τη θητεία η διαδικασία. Ωστόσο δεν είχαμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε περαιτέρω τα θέματα και επομένως καλύτερα είναι να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια αυτή. Και στην τελευταία συνάντηση των Προέδρων των επιτροπών ε, διαπιστώθηκε τροποποίηση της θέσης. Εγώ ήξερα από την αρχή ότι υπάρχουν αντιθέσεις ε, όσον αφορά τις απόψεις. Στο σεμινάριο του προηγουμένου Φεβρουαρίου μερικοί ήθελαν κατάργηση του άρθρου 50, άλλοι ήθελαν να παραμείνουν όσα είχαν τα πράγματα. Ε, είχε, είχαμε προωθήσει μία πρόταση συμβιβαστική, αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι πρόεδροι επιτροπών το ξανασκέφτηκαν το πράγμα και άλλωστε δεν είναι τόσο ζωτικό το θέμα, δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι κρίμα βέβαια που ε, μετά από πέντε χρόνια θητείας ε, και μετά από ε, την εμπειρία και τη σοφία την οποία έχουμε συλλέξει αυτά τα πέντε χρόνια δεν είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τα πράγματα γιατί σίγουρα η επόμενη θητεία δεν θα έχει μεγάλη εμπειρία εξ αρχής αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Η κυρία Γιαννάκου δεν έχει έρθει ακόμα. Να περιμένουμε ακόμα πέντε λεπτάκια. Η παρέμβασή μου για τα άρθρα 49 και 50 στην ουσία ε, ολοκληρώνει και την εξέταση του άρθρου 10 της ημερησίας διάταξης. γιατί είχαμε προβλέψει συζήτηση του εν λόγω θέματος Α, ο κύριος Μέσερ Σμιτ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Για το σημείο 10 πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδε στη διάσκεψη των Προέδρων είχαμε μια συζήτηση για τι διεργασίε για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση διαδικαστικά και ο κύριος Σούλτς είχε προναγγείλει διάφορες δυνατότητες εναλλακτικέ που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Τις εξετάζουν οι ομάδες τώρα. Ένα πράγμα όμως όπου φαίνεται ότι υπήρξε συνένεση είναι η ανάγκη διευρυμένης ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα μέλη ή μη μέλη, μη, μη μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών όταν έχουμε τέτοιες συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε πρώτη ανάγνωση συμφωνίες όπως γνωρίζετε τα μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογία στην Ολομέλεια στο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, διότι αν κάτι τέτοιο εγκριθεί τότε καταπίπτει μια τέτοια συμφωνία πρώτη ανάγνωση. Είναι σημαντικό λοιπόν μέλη, μη μέλη τη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που θέλουν να επηρεάσουν τι διεργασίε να υποβάλουν τι τροπολογίε του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη τα οποία δεν είναι μέλη τη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό, αν όχι στην έκθεση, στην ανακοίνωση των Προέδρων Βουλευτών Επιτροπών Οτών, κ. Κασίνη, προσέθη σε αυτή τη συνάντηση για αυτή την αναγκαιότητα. Καλό θα ήταν να δούμε μια τέτοια δυνατότητα να τροποποιήσουμε τα πράγματα όταν έχουμε τέτοιου είδου συμφωνίε πρώτη ανάγνωση υπό εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σημειώνω αυτά που είπατε. Θα δούμε στην επόμενη συνάντηση και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Ωραία. Ο κύριο Νταφ. Νομίζω ας να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, πρόεδρε. Για την έκθεση για τα εθνικά κοινοβούλια και να επανέλθουμε στο θέμα του καθεστώτος των πολιτικών κομμάτων όταν έρθει η κυρία Γιαννάκου. Μου λένε ότι η κυρία Γιαννάκου έρχεται. Είναι σκόπιμο να την περιμένουμε. Posso soltanto introdurla. Ah, Hefner, ναι, ναι. prego. Ο Χέφνερ. Θα ήθελα σύντομα μόνο να εκμεταλλευτούμε το χρόνο ώστε να γνωστοποιήσω στα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής τη συζήτηση των συντονιστών σήμερα ότι εγώ στο σημείο εκείνο όπου εμείς κάνουμε λόγο για μια γνωμοδότηση, μια μελέτη της ε, νομικής υπηρεσίας μας για το θέμα το οποίο από την Επιτροπή Αναφορών μας είχε διαβιβαστεί σε μας σε σχέση με πιθανή προσπάθεια ανεξαρτοποίησης ε, ε, κρατών ή ε, μημάτων κρατών της Ευρώπης ε, ο πρόεδρος να μην δώσει την έγκρισή του να συνταχθεί μια τέτοια γνωμοδότηση. Και αυτό με ξενίζει, με ξενίζει μια και πιστεύω ότι όταν μια κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου διακομματικά εκφράζεται υπέρ μια τέτοια γνωμοδότηση ή μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είναι δυνατό να συνταχθεί μια τέτοια μελέτη και να μην τροχοπεδηθεί εκ των άνω. Ε, κατά τα άλλα όμως πιστεύω ότι με τις ψηφοφορίες, με τη σειρά που προβλέπετε μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσουμε με το σημείο της κυρίας Γιαννάκου, αλλά να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι άλλο για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Δεν προβλέπουμε μόνο ψηφοφορία, αλλά και συζήτηση. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες είναι σωστό να δώσουμε χρόνο στην συζήτηση. Ε, εγώ είχα πει ότι είμαι έτοιμος, ήμουν έτοιμος να αντικαταστήσω την κυρία Γιαννάκου, αλλά μου λένε ότι έρχεται. Έρχεται πρόεδρε, να Πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Γιαννάκου να θυμίσω ότι με επιστολή στις 5 Μαρτίου ο πρόεδρος της ΚΟΡΕΠΕΡ, ο κύριος Σωτηρόπουλος, ενημέρωσε για το σχέδιο πακέτου συνολικού συμβασμού που συμφωνήθηκε στην ΚΟΡΕΠΕΡ την ίδια μέρα. Πήρατε το έγγραφο αυτό αυτή την εβδομάδα και γνωρίζετε ότι από την έκτακτη συνάντησή μας ε, στην προηγούμενη Δευτέρα. Η κυρία για να ενημέρωσε για την επιτυχία του τριλόγου στις 25 Φεβρουαρίου, όπου κατά βάση έγιναν δεκ... έφτασε η κυρία Γιαννάκου, έγιναν δεκτά έλεγα κάποια από τα αιτήματά μας. Άρα στη φάση αυτή θα σταματήσω και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γιαννάκου, για να μας παρουσιάσει την τελική έκβαση του τριλόγου και το, το πλαίσιο που πετύχαμε σαν διαπραγμάτευση του πλευράς και κοινοβουλίου. Κύριε Γιαννάκου. Πρόεδρε, ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και σας προσωπικά ε, για την βοήθεια την οποία παρήχατε και για την ε, ουσιαστική συνεννόηση η οποία υπήρξε μεταξύ μας και που μας οδήγησε σε ευτυχή κατάληξη κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Είναι γεγονός ότι η έκθεση αυτή και ιδίως η έννοια του στάτους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων δημιούργησε πολλές ανησυχίες στα κράτη-μέλη και πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό και καθυστέρησε ο Τρίλογος. Όπως αντιλαμβάνεστε ε, υπήρχαν και προεδρίες που δεν μπορούσαν να επιβάλλουν μια ενιαία γραμμή στο Συμβούλιο και σας υπενθυμίζω κύριε Πρόεδρε ότι στο τέλος επί ελληνικής προεδρίας δόθηκε εντολή συνολικής διαπραγμάτευσης διότι σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα ήταν πολύ δύσκολο να γίνεται επιμέρους διαπραγμάτευση και να μην έχει την εντολή η Προεδρία του Συμβουλίου για συνολική διαπραγμάτευση. Κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησής μας, στην προηγου... όχι στην προηγούμενη, στην αμέσως προηγούμενη, ε, Ολομέλεια του Στρασβούργου στη συνάντηση που είχαμε με την Προεδρία και τον Επίτροπο τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς ε, επετεύχθη συμφωνία τελικά μεταξύ των τριών πλευρών ε, η οποία μπορεί να μην ήταν μέσα στο πλαίσιο απόλυτα της δικής μας άποψης της αρχικής αλλά ωστόσο δεν ήταν απομεμακρυσμένη η συμφωνία που επετεύχθη από τους στόχους που είχαμε από την αρχή. Δηλαδή θέλαμε την ανεξαρτησία α, της α, εγγραφής χωρίς πολιτική παρέμβαση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, δεν θέλαμε περισσότερα χρήματα για τα κόμματα και το είχαμε τονίσει και το είχαμε πει προς πάσα κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους ε, θέλαμε να υπάρχει πραγματικό νομικό στάτους σε όλες τις χώρες να γίνει αποδεκτή η άποψή μας ε, τα, οι πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να γίνονται κατευθείαν μέλη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θέλαμε να ρυθμιστούν ζητήματα που είχαν σχέση ε, με την αύξηση της προσωπικής συνεισφοράς ιδιωτών στα κόμματα ζητήματα που είχαν σχέση με τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα αλλά και τα κόμματα ως προς το carry-over, τη μεταφορά δηλαδή κεφαλαίων για την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά τα ζητήματα ρυθμίστηκαν ευμενώς σε σχέση με την άποψη που είχαμε εμείς από την αρχή και αυτή την ώρα τελειώνει και η υπόθεση της έκθεσης που έχει το, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η έκθεση κυρίας Κρέσλε, ε, για το καθαυτό funding και τις κυρώσεις στην περίπτωση που παρατηρούνται ε, ζητήματα που δεν εναρμονίζονται με τον κανονισμό. Ε, απ' την άλλη πλευρά κύριε Πρόεδρε παρά τη δική μας άποψη ότι το ρεζίστρι για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έπρεπε να είναι μια απλή υπηρεσία του Κοινοβουλίου τελικώς επελέγει η λύση ενός ανεξάρτητου φορέα κατά κάποιο τρόπο μέσα στο Κοινοβούλιο μιας ανάνς θέση του Συμβουλίου την οποία αποδεχθήκαμε γιατί αποτελούσε επιμονή όλων των μερών που απαρτίζουν το Συμβούλιο. Αυτό που είναι σημαντικό κύριε Πρόεδρε είναι ότι προβλέπεται στον κανονισμό ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού αφενός ε, και αφετέρου προβλέπονται ανάλογες εκθέσεις από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ε, πρώτων εκλογών του 2019 έτσι ώστε να ε, παρακολουθηθεί το πώς πάνε τα κόμματα αν ε, ο κανονισμός αυτός έχει εξαντλήσει τη δυνατότητά του να προσφέρει όσα από την αρχή είχαν προβλεφθεί και βέβαια κύριε Πρόεδρε ο δρόμος είναι ανοιχτός κάθε φορά για να διορθωθούν στο μέλλον ε, πιθανά λάθη, πιθανές αυλεψίες κτλ. Ε, έχει τεράστια πολιτική σημασία το ότι έληξε ο τρίλογος αυτός καλά υπό την έννοια ότι ήδη τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν προτείνει και τους υποψηφίους τους για, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρά το γεγονός ότι δεν θα αρχίσει αμέσως να εφαρμόζεται ε, διότι ε, λογικά πρέπει πλήρως να εφαρμοστεί την 1η Πρώτου του 2017. Πρέπει να δοθεί χρόνος δηλαδή στα κόμματα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στη νέα πραγματικότητα. Να επιλέξουν πιθανόν ε, οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης για να εγκατασταθούν και ούτω καθεξής. επομένως προσλαμβάνει και μια άλλη πολιτική διάσταση το γεγονός ότι πια έχει ληφθεί η απόφαση να μην είναι διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις τα κόμματα αλλά να έχουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό στάτους και να ανταποκρίνονται σε αυτό που προβλέπει η συνθήκη. Διότι είναι σημαντικό το άρθρο της συνθήκης με τις συγκεκριμένες προβλέψεις του. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και πάλι τη διαπραγματευτική ομάδα και όλους, όλα τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν και τους συντονιστές τους και τους ε, σκιώδεις εισηγητές αλλά επαναλαμβάνω και εσάς προσωπικά διότι η Επιτροπή δούλεψε ε, με σωστό και ε, πολύ συνεργάσιμο μεταξύ των μελών τρόπο και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφισή του θα πάει τον Απρίλιο στην Ολομέλεια άλλωστε έτσι είχε προβλεφθεί και από την αρχή και αμέσως μετά θα το υιοθετήσει το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι θα είμαστε και συνεπείς στο στόχο μας και στις διακηρύξεις μας πρώτων εκλογών να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση ε, η οποία να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη συνεργασία και όλη την ε, βοήθεια και την προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της ε, δουλειάς που κάναμε που ε, τράβηξε αρκετά. Δηλαδή διατέθηκε πολύς χρόνος, πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά και με ευτυχή αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία όμως ζήτησε να πάρει τον λόγο ο κύριος Φόξ. δώσω τα 10 λεπτά στην κυρία Γιαννάκου για να μας πει πόσο καλά είναι όλα αυτά. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι η συμφωνία είναι πολύ κακή, είναι bad deal. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προ... υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ε, πρόκειται για χρηματοδότηση η οποία ε, παίρνει λεφτά από τον ε, Ευρωπαίο φορολογούμενο και τα δίνει σε αυτά τα κόμματα. Απ' την άλλη πλευρά όμως ίσως και ακόμα πιο σημαντικό ε, δίνει χρήματα σε σχέση με το κατά πόσον συμφωνούμε με τις αξίες τους, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία. Φανταστείτε, φανταστείτε στην, στην εθνική πραγματικότητα, στα εθνικά κοινοβούλια, να πούν η πλειοψηφία των βουλευτών δεν συμφωνούμε με τις αξίες του τάδε κόμματος, του παίρνουμε τη χρηματοδότησή του πίσω. Ε, ε, υπάρχουν ας πούμε ο συνάδελφος Μποντ ε, εδώ ο οποίος έχει εκλεγεί με ένα κόμμα το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Αλλά τι θα γίνει, θα του αρνηθούμε του κόμματος αυτού την χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς τα κόμματα με τα οποία δεν συμφωνεί είναι μέσω της εκλογικής διαδικασίας και μέσω των καλπών. Αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία. Ευχαριστώ κύριος Μπροντ. Είναι αναμφισβήτητο ότι η ε, ε, το δικαίωμα του ε, συναθρίζεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει κανείς να επιτρέψει είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με κάποιες απόψεις την δυνατότητα όλων των πολιτικών και όλων των κομμάτων να εκφράζουν τις απόψεις τους και βεβαίως κατά αυτή την έννοια θα πρέπει η πολιτική τάξη να ακολουθεί τις αρχές τις οποίες έχει ε, επί τον οποίο έχει συμφωνήσει. Ε, από την άλλη πλευρά ε, μην λησμονούμε ότι αυτές οι ελευθερίες της έκφρασης και του συναθρίζεστε είναι αρχές οι οποίες διέπουν και τα ευρωπαϊκά κόμματα. Υπάρχουν και άλλες αρχές, ας πούμε, της μη διακριτικής μεταχείρισης είναι λίγο πιο υποκειμενικές. Έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες γιατί ήδη οι πρώτες προσπάθειες να απαγορευτεί η καταγραφή πολιτικών σχηματισμών έγινε χωρίς αναφορά ε, στον ε, λόγο για τον οποίο ε, δεν μπορεί να γίνει η καταγραφή του. Είναι δηλαδή σαν να κατηγορείς κάποιον χωρίς να του απαγγέλει συγκεκριμένη κατηγορία. Ο κύριος Ντάφ. Πρόεδρε, η ομάδα των φιλελευθέρων υποστηρίζει στεναρά την συνενετική θέση που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτριά μας κυρία Γιαννάκου για την αντοχή της και συνέχεια με σθένος που έδωσε σε αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο. Η συμφωνία θα αναβαθμίσει το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουν να μετεξελιχθούν σε αξιόπιστα, σύνθετα πολιτικά μορφώματα ως κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επίπεδο εκείνο στο οποίο, το οποίο χρειάζεται η δημοκρατία μας να λειτουργήσουν. Η διεργασία αδιαγραφής είναι μεγάλη πρόοδος σε σχέση με το σύστημα. Συνεισφέρει στη διαφάνεια και εμπλέκει και το Συμβούλιο, καθώς επίσης και το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε και τα δύο σώματα από πλευράς νομοθετικής αρμοδιότητας να εμπλέκονται. Και δεν είναι μια, ας το πούμε, ασίδωτη συμφωνία όπου κομματικοί εκπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούν να καταδιώκουν πολιτικές ομάδες που δεν, τους, ε, που δεν είναι της αρεσκίας τους. Ε, αρχές και αξίες ε, που όλοι υποχρεούνται να σέβονται φυσικά είναι εκείνες που θεσπίζονται και εκφράζονται στην συνθήκη και στην χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τα άλλα η ρήτρα αναθεώρησης ε, όπως η ίδια η συγγήτρια ανέφερε είναι σημαντικό στοιχείο και αυτή και γοργά θα συναγάγουμε βιωματικά από την πρακτική εφαρμογή εμπειρικά τα σωστά συμπεράσματα και θα δοθεί η συνέχεια σε αυτό το νομοθέτημα όπως θα πρέπει ώστε για το 2019 στις ευρωεκλογές να ισχύουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ζήτησαν πολύ το λόγο να, να είστε πιο σύντομοι. Ο κ. Στάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να ε, ενοχλήσω συναδέλφους. θέλω να πω κάτι για να μην έχω βάρο στην καρδιά μου. Κατά την άποψή μου σήμερα τα πολιτικά κόμματα είναι υπερβολικά ογκώδεις οργανώσεις. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται μόνο από τις συνδρομές των μελών τους. Έχουν μέλη, τα μέλη αποφασίζουν πόσα χρήματα θα δωρήσουν σε μια πολιτική ε, σε ένα πολιτικό στόχο. Η έκθεση λοιπόν θα έπρεπε να πει δεν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση από επιχειρήσεις, από λόμπι, από παρατρεχάμενους εν γέννη και κατάργηση της χρηματοδότησης των πολιτικών οργανώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, μόνο από τις συνδρομές των μελών. Ξέρω τι πρέπει να κάνετε τώρα, ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε ξανά ωστόσο στην επόμενη θητεία. Διότι ως πολιτικά, τι κάνουμε ως πολιτικά κόμματα με τα χρήματα που μας δίνουν οι φορολογούμενοι και τα επιπλέον χρήματα που παίρνουμε με όχι μεγάλη διαφάνεια από άλλους οργανισμούς. Χαζές διαφημίσεις στην τηλεόραση, ε, κολλάμε αφήσει στις πόλεις μας με τις φωτογραφίες μας, προσλαμβάνουμε προσωπικό. Αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικά επίφοβο. Τέλος πάντων θα, ψηφίσω την ε, συνένεση σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άναν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Τόμας Τζέβερσον δυστυχώς δεν είναι μέλος της επιτροπής μας. Ο τρίτος πρόεδρος τον είπα ωστόσο είχε πει κάτι ότι το να υποχρεώσουμε κάποιον να παράσχει πόρους για ιδέες που δεν πιστεύει είναι αμαρτωλό και τυραννικό, είπε ο Τζέφερσον. Ο κύριος Χέφνερ. Θα ήθελα μόνο σύντομα για την δική μου πολιτική ομάδα να πω ότι εμείς σε εκτενείς και κοπιώδεις διαβουλεύσεις αυτό το συμβιβασμό τον οποίο επετέφθη τον υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Χρειάζεται η δημοκρατία πολιτικά κόμματα και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα ποια κόμματα προσπαθούν να κερδίσουν την ψήφο των πολιτών δεν θα πρέπει αποκλειστικά να κρίνεται από την οικονομική ισχύ και δύναμη που συλλέγουν τέτοιου είδους κόμματα. Είναι πολιτιστική και πολιτισμική πρόοδος να αναζητούνται τρόποι και να εξευρίσκονται τρόποι και δυνατότητες ώστε όλοι να έχουν το δυνατόν ίση πρόσβαση σε τέτοιες πηγές. Θα ήθελα πριν από την ψηφοφορία να πω το εξής. Απόλυτα μπορώ να κατανοήσω ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων που θα τεθούν σε ψήφιση. Αλλά αναμένεται, πιστεύω από κάθε Ευρωβουλευτή και πρέπει να αναμένεται, ότι για τις προτάσεις που εδώ υποβάλλονται προς ψήφιση τις γνωρίζει και προτού ψηφίσει η μιλήση να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό πολύ σύντομα στον κύριο Μπρόνς. Κύριε Μπρόνς είπατε ότι θα καταψηφίσετε, διότι αν υπερψηφίζατε αυτή την πρόταση τότε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να αποφασίζει ποια κόμματα θα ενέκρινε και ποια όχι, κατά το δοκούν ασίδωτα, με προσωπικά ίσως κριτήρια. Και γι' αυτό είπατε θα καταψηφίσετε αυτή την έκθεση και κατά του status quo. Ένα πράγμα μας να σας πω επ' αυτού. Σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία είχαμε μια διαδικασία όπου μια πολιτική ομάδα αυτού του σώματος συνέλεξε υπογραφές ώστε κάποια πολιτικά κόμματα να μην έχουν άδεια να λειτουργούν. Αυτό είναι το status quo. Αυτή είναι η διαδικασία όπως ισχύει. Τώρα έχουμε μια νέα διαδικασία που βρήκαμε, που αυτό να το καθιστά αδύνατον βρήκαμε ένα μηχανισμό που καθιστά ανέφικτο και αδύνατο για πολιτικούς λόγους ευρωβουλευτές ή μια πλειοψηφία ευρωβουλευτών απλά και μόνο να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει κόμματα ή να τα απαγορεύει ώστε αυτό να γίνεται από ένα ανεξάρτητο σώμα, ένα ανεξάρτητο φορέα από ένα σώμα το οποίο θα συναπαρτίζεται από ανεξάρτητες προσωπικότητες μη εμπλεκόμενες και ουδέτερες, αμερόληπτες, ώστε στο τέλος να είναι μια απόφαση που από κοινού θα πρέπει να εγκρίνουν το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να ασκείται προσφυγή σε δικαστήριο κτλ. Βρήκαμε ένα σύνθετο μηχανισμό που ακριβώς αυτό οδηγεί στο να αποφεύγεται αυτό το οποίο εσείς ισχυριστήκατε ότι θα γινότανε. Αν ουσιαστικά τα εννοείτε όλα αυτά σοβαρά θα έπρεπε να υπερψηφίσετε αυτό το συμβιβασμό όπως όλοι θα κάνουμε. Και που όλοι έχουν συμμετάσχει έντονα σε αυτό σε, διαφορά, σε διαφορά και αντιδιαστολή με εσά κύριε Μπρόνς. Ευχαριστώ κύριος Γκουαλτιέρη Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω απλά να εκφράσω την βαθιά υποστήριξη της σοσιαλιστικής ε, ομάδας στο συμβιβαστικό κείμενο για το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλη την διαπραγματευτική ομάδα. Γνωρίζουμε ότι είναι συμβιβασμός, θεωρούμε παρά τα αυτά ότι ο συμβιβασμός αυτός είναι καλός, που επιτρέπει να προχωρήσουμε ουσιαστικά προς τα μπροστά και πολιτικά και θεσμικά και συνταγματικά δίνοντας ένα νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ακριβώς ε, επιβάλλουν και οι συνθήκες που, αναφέρουν, που αναθέτουν στα πολιτικά κόμματα την ευθύνη να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής συνείδησης της Ευρώπης και την έκφραση της Βούλης των Πολιτών της Ένωσης. Η έκθεση αυτή αποτελεί μια σημαντική ψηφίδα στην κατα στη δημιουργία μιας πολιτι... πιο πολιτικής και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορεί να στηριχθεί σε ένα πολιτικό χώρο που θα είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκό. Σε ό,τι αφορά τι ανησυχίε που εκφράστηκαν, ο κύριος Χέφνερ διευκρίνησε ήδη ότι ο κανονισμός αυτός ενισχύει το σύστημα των εγγύσεων για την ελευθερία έκφρασης γνώμης των πολιτικών κομμάτων, καθιστά πιο σύνθετη δηλαδή την διαδικασία ελέγχου του σεβασμού των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και της, διαγραφή, και της καταχώρησης και διαγραφής. Είναι ένα κείμενο λοιπόν που προσφέρει εγγυήσεις, είναι σημαντικό κείμενο, θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ νωρίτερα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί κάναμε αυτό το σημαντικό βήμα μπρο στην ενεργοποίηση των αρχών της συνθήκης. Ο κύριος Μπρόντς έχει το λόγο. Όχι, ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Μπρόντς μίλησε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω εξ ονόματος Ενωτικής Αριστεράς να πω ότι υποστηρίζουμε αυτό το συμβιβασμό που πετεύθη. Ήταν μια έντονη σε βάθος εργασία επί μεγάλο πολιετές χρονικό διάστημα και ίσως μια ένταση της συζήτησης ακριβώς για τα διαφορετικά προβλήματα που εξακολουθούν να έχουν κάποιοι ευρωβουλευτές, κάποια ε, κοινοβουλευτικά κόμματα, κάποιες κοινοβουλευτικές ομάδες ε, αν έχουν τέτοια προβλήματα, να μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε ένα ταχύτερο αποτέλεσμα. Βλέποντας το εύρος, την εμβέλεια, την ευθύνη που με αυτό το χαρτοφυλάκιο καταφέραμε να ρυθμίσουμε και να έχουμε συνειδητοποιήσει, Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους συναδέλφους για το ότι στο τέλος τέλος καταλήξαμε σε συμβιβασμό στον τριμερή διάλογο που λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και των κρατών μελών όσον αφορά τον ρόλο της ε, συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων στη δημοκρατική διαμόρφωση των πραγμάτων και των απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο με αυτόν τον τρόπο όπως ρυθμίστηκε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι εδώ αναφερόμαστε στη δραστηριότητα και των πολιτικών κομμάτων και συνδέουμε αυτή τη δραστηριότητα στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δηλαδή στη δημοκρατική εκείνη, στο δημοκρατικό υπόβαθρο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι ένα δημοκρατικό πλαίσιο εργασίας ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να απλουστεύεται από ό,τι σε σχέση με το status quo. Είναι λοιπόν ο συμβασμός ένα σωστό βήμα, ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ο Μέσερ Σμιτ παρακαλώ. Ο κύριος Ντάφ είπε ότι ε, τα ισχυρά φεντεραλιστικά κόμματα είναι αυτά που χρειάζεται η δημοκρατία. Θα μπορούσα να συμφωνήσω κύριε ε, Ντάφ, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι η δημοκρατία χρειάζεται κυρίως αμοιβαία εμπιστοσύνη, ε, χρειάζεται κοινή γλώσσα. Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτό χρειάζεται η δημοκρατία. Τώρα, μπορεί κανείς να πάει στην ε, Grand Place εδώ στις Βρυξέλλες ή στην Piccadilly Square στο ε, Λονδίνο ε, και να μιλήσει για την, εκεί για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και να τους πει ότι αν πιστεύουν, να τους ρωτήσει αν πιστεύουν ότι τα φιντελιστικά κόμματα θα σώσουν την Ευρώπη να δούμε αν θα απαντήσει κανείς θετικά. Ευχαριστώ κύριο Σόφλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχικά δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο γιατί νομίζω ότι εδώ γίνεται κανονική συζήτηση και ήθελα και εγώ να κάνω τη μικρή μου σύμβολη. Ε, όπως και άλλοι προηγούμενοι ομιλητές, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γιαννάκου. Συζητάμε εδώ και πολύ καιρό το θέμα αυτό και νομίζω ότι η δουλειά που έκανε είναι εξαίρετη. Ένα ουσιαστικό σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω, επί της ουσίας δηλαδή, είναι ότι η πραγματικότητα ε, ορίζει το πολιτικό πεδίο. Ωστόσο, ε, πρέπει να πούμε ότι ε, δεν έχουμε εδώ ιδεολογική συζήτηση. Ε, πρέπει να κάνουμε μια ορθολογική πραγματιστική συζήτηση. θα Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να γίνει διαφανής και λογική μια κατάσταση που οπωσδήποτε θα υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει να απαντήσει η κυρία, κυρία Γιαννάκου. Θέλετε να απαντήσετε, θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε να απαντήσετε, θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητο. Κύριε Πρόεδρε, το μόνο που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους και να σημειώσω ε, ότι η αποδοχή από τα κόμματα των αρχών και των αξιών της Ένωσης δεν είναι οποιονδήποτε αρχών και αξιών. Είναι των αρχών και αξιών που περιγράφονται στη συνθήκη. Και δεν τίθεται θέμα να μην γίνονται σεβαστές αυτές, και οι, αυτές οι αρχές και οι αξίες. Δεν μιλάμε λοιπόν γενικός και αορίστος για τις πολιτικές απόψεις του κάθε κόμματος, μιλάμε για τον σεβασμό των αρχών και αξιών που περιγράφονται και όπως περιγράφονται στη συνθήκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και δίκαιο και έντιμο ώστε κάποιος που χρηματοδοτείται και τελεί υπό τους κανόνες να σέβεται. Επομένως δεν έχουμε θέμα όπως περιγράφει προηγουμένως ότι αυτό αποτελεί απόκληση και αυτό που είπε ο κύριος Φόξ και τα λοιπά. Και πρέπει να σας πω ότι στο επίπεδο του Συμβουλίου αυτά όλα έγιναν αποδεκτά από όλους. Ε, σας ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε ε, στην ψηφοφορία. Μία ψήφος διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 18 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά, μία αποχή και επομένως εγκρίνεται η έκθεση. Θα ήθελα να συγχαρώ για μια ακόμα φορά τη συνάδελφο κυρία Γιαννάκου και να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα της πρόκλησης της Ευρώπης ε, γιατί θέλουμε πραγματικά να οδηγηθούμε προς την Ενωμένη Ευρώπη. Επομένως, ε, εκφράζω την ε, χαρά μου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1, ε, Ραμόν Τρεμόζα, δεν ε, γίνεται δεκτή. Ε, γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί του τίτλου. Δεν έχουμε ε, άδεια για κάτι τέτοιο. Η άδειά μα ε, ήταν για συγκεκριμένο τίτλο. Επομένως, τροπολογία 82, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 83, Άντριου Ντάφ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 Ντάφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Α υπέρ κατά αποχές μία αποχή εγκρίνεται και περνάμε επομένως απευθείας Στην τροπολογία 88, Γκουαρτιέρη και Ριπών, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Β, υπέρ. Θέλετε να μιλήσετε κύριε Ντάφ. Κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί μετά από τη συζήτηση στην ε, Επιτροπή ε, ενστερνιστήκατε την ουσία της ε, τροπολογίας μου. Ωστόσο, η αγγλική διατύπωση στο συμβιβασμό θα πρέπει να λέει commend national parliaments for taking steps to. Αυτή είναι η, σωστή από γραμματικής απόψεως διατύπωση, αλλά και από πολιτικής απόψεως. Αυτή είναι η βέλτιστη στην αγγλική διατύπωση. Σας ευχαριστώ. Ωστόσο, το κείμενο το οποίο εγώ θέλω να προτείνω λέει ακριβώς αυτό. Ε, συνστήνει τα εθνικά κοινοβούλια να πάρουν μέτρα κτλ. Ίσως, το, ίσως κάποιο πρόβλημα έχει το, η αγγλική διατύπωση. Διαβάζω στα Ιταλικά λοιπόν. Συστήνει τα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν, ε, να λάβουν μέτρα ώστε. Ο Ναι, αλλά η τροπολογία μου λέει commands. Όχι recommends, commands. Ε, αυτό σημαίνει ότι συγχαίρει τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια διότι έχουν αναλάβει ε, ε, έχουν ξεκινήσει βήματα προς. Είναι, είναι πιο ενθαρρυντική διατύπωση κατά την άποψή μου. Να σας πω ότι το πρόβλημα είναι γλωσσικό. Εσείς ε, διαβάζατε στα αγγλικά το κείμενό σας και οι διερμηνείς μου λέγανε συστήνει ε, να πούμε εκφράζει την ικανοποίησή του. Comments και όχι comments. Με αυτή τη γλωσσική διόρθωση δεν έχω πρόβλημα. Allora, pongo in votazione l'emendamento di Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ, Β, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε. Τροπολογία 98, Γκουαλτιέρη και λοιπόν, υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Δεκτό. 99 υπολογία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα προχωρούμε στην τροπολογία Ε. Όχι. Διορθώνει ο πρόεδρος. 103 Μπασέσκου υπέρ. Τροπολογία 103. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το 104 έχει καταπέσει. Συμβαστική Ι. Ε. Υπέρ. κατά εγκρίνεται να σας πω την αλήθεια αλλά ας κάνουμε και ηλεκτρονικό έλεγχο ψηφίζουμε την συμβιβαστική E ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία Τροπολογία 109. Μέσα Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Σίγματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Ζ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προχωράμε. Τροπολογία 115 Fox υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 Fox υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 Γκουαλτιέρη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 120 Φόξ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, του Ρανζέλ υπέρ. Να μετρήσουμε. Ηλεκτρονικά καλύτερα. Για την 122 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για μια ψήφο. Τροπολογία 123 υπέρ. 123 Ραντζέλ υπέρ, κατά, πάλι θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 123 Ρανζέλ. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάλι για μια ψήφο. 124 ε, Fox, favorevoli. 124 Fox υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 125 και 126, ημένα 125 του Σόλτση, 126 του Γκουαλτιέρη και λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127, Νταφ, Κλάις, Γκουαλτιέρη, Είναι πολλέ ίδιε τροπολογίε από 127 έω 130 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία H. Ήτα. Εδώ έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμηματο Κατά. αποχε Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά εγκρίνεται νομίζω αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο για το δεύτερο τμήμα Τη συμβαστική ή έρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 13 προς 11 αυτό σημαίνει ότι Καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στην 137. Γκουαλτιέρη και λοιπή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139. Όχι. Ναι. Πρέπει να ψηφίσουμε. Όχι. Bisogna votarlo, sì sì, perché è stato respinto. 139. 139 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 140. Χέφνερ. Και Τάραντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 και 42 και 43. Υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψηφίσετε όλοι. Απορρίπτεται. 10 προς 14.

αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, παρακαλώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι απορρίφθηκε η 147, μπορούμε να το ελέγξουμε. 147. Εγώ νομίζω ότι είχε απορριφθεί, λέει ο πρόεδρος, και άνετα Μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο στην 147. Ψηφίζουμε μαζί την 146 και την 147, γιατί είναι όμοιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Συμβιβαστική I, φίτα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγώ θα έλεγα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα του ΆΗ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα δεν υπάρχει πια. Πρέπει να δούμε βέβαια τι δεν έχει καταπέσει τώρα έτσι όπως έγινε. Η 149 κατέπεσε. Συμβιβαστική L. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Έχει καταπέσει 152. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε και πηγαίνουμε στην 159 τροπολογία Σόλτς υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε θέλετε να κάνουμε έναν έλεγχο ωραία ψηφίζουμε για την 159 Σόλτς ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 9 προς 14, 159, 160 υπέρ, κατά, η ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 160. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 161 162 και 163 είναι οι ίδιες, ψηφίζουμε την 162-163. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 162 και 163. Ψηφίζουμε τις τροπολογίε 164, 165, 166. Υπέρ να παρακαλώ σηκώσετε το χέρι σας. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 έχει καταπέσει γιατί εγκρίθηκε 166 168, 69, 70, 71 και 72 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζονται από κοινού υπέρ, κατά εγκρίνονται Ψηφίζουμε την τροπολογία 173 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174. Όχι, μισό. Έχουν εγκριθεί 178-172, άρα έχουν καταπέσει. Από την 174 μέχρι την 179 έχουν καταπέσει διότι εγκρίθηκαν οι 168-172. Ψηφίζουμε την 180 τροπολογία υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ας γίνει ένας έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική εν, νη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στην συμβιβαστική 183 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε 184, 85, 86, 87 και 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Τροπολογία 190, Ashley Fox, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. ψηφίζουμε το συμβιβασμό OUR κατά τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται. Όχι, είμαι σίγουρος ότι εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά καλύτερα σε αυτή την περίπτωση να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί του δευτέρου τμήματος ε, του συμβιβασμού O. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Όντως απερίφθη. Αυτό σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε την 197 υπέρ κατά δύσκολο να αξιολογήσω το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, μία με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. Τροπολογία. Τροπολογία 199. <coughs> συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 198 δεν ψηφίζουμε. Α, όχι, είναι συμβατό. Επομένως ψηφίζουμε και την τροπολογία 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 198 Ashley Fox. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 201, 202, 203 καταπίπτουν. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, έκανα λάθος. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 201, 202, αλλά ψηφίζουμε τη 203, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 204, και μαζί η τροπολογία 205 γιατί είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207, όχι λέει ο Πρόεδρος, έχει καταπέσει το ίδιο και 206. Το ίδιο και 206. Φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 2. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Μάλλον όχι. Επί του 12 τροπολογίες 5 και 6 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. Τροπολογία η τροπολογία 7 ήδη ε, περιέχεται στην τροπολογία 4, αλλά δεν ψηφίζουμε. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 9 και 10 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται, ναι. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 και 13 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 φόξ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 και 16 ταυτόσημες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 17, Fox, υπέρ. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Τι κάνουμε, ναι, ψηφίζουμε τη 17 Fox υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. πίπτη Φτάσαμε στο συμβιβασμό π. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός, μάλλον όχι, τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Q. Κατά τμήματα θα ψηφίσουμε, ρωτάει ο πρόεδρος. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. Καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβιβασμός Q, δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όντως απερίφθη. Έχω μια υποψία, λέει ο Πρόεδρος, ότι δεν λειτουργεί η δικιά μου η κάρτα. Α, δεν είναι κάτι. Ε, Va bene, va bene. Allora, eh, siamo all'emendamento 24. Πού είμαστε? Τροπολογία 24 έχει καταπέσει. Τροπολογία 25, 26, 28. Λοιπόν, φτάνουμε στο συμβασμό R. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική δεν είμαι βέβαιος. Συμβιβασμός R. Λοιπόν, από την αρχή προσπαθούσα να ψηφίσω και προφανώς δεν ψήφιζα. Κάποιο πρόβλημα είχε η κάρτα μου, λέει ο Πρόεδρος. Πέρα τη ψηφοφορία, ό,τι έγινε έγινε τώρα, η ψήφιος μου προφανώς δεν προσμετρήθηκε πουθενά. Εν πάση περιπτώσει ο συμβασμός αυτός απορρίπτεται για μία ψήφο. Επομένως, πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 29 και την τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε επαλήθευση. Ας την κάνουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Καταπίπτει. Συμβιβασμός S. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι πάμε απευθείας να ψηφίσουμε το επόμενο συμβασμό που είναι ο συμβασμός T. Υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 12 ψήφοι πέρα, 11 κατά. Φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβασμός U υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία για το συμβιβασμό U Πέρας. Απερίφθη. Επομένως ψηφίζουμε τις τροπολογίες 44, 45 και 46. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Άρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 50 υπέρ ακόμα και αν εγκριθεί η τροπολογία, τότε, ε, είναι, τότε καταπίπτει, όχι μόνο, εάν, ε, όχι μόνο σε σχέση με, την, ε, με το συμβασμό. Καταπίπτει έτσι κι αλλιώς. Προχωρούμε λοιπόν. Τροπολογία 52 υπέρ. κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν επί της τροπολογίας 52 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έσφαλα. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε απευθείας λοιπόν στην τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρο... Συμβιβασμός W κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60, 61, 62, 63, 64 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 65 και 66 που είναι ταυτόσιμε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67, 68. Ταυτόσιμες επίσης. Τις ψηφίζουμε. 66-67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως, τροπολογία 69 καταπίπτει. Τροπολογία 70, Fox. Κατά αποχές να κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 70 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται το 70 τροπολογία 70 κατέπεσε η 72 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συγγνώμη πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω γιατί η 71 θεωρείται ότι κατέπεσε εφόσον εγκρίθηκε η 70. Προτείνουν διαφορετικά κείμενα, δεν είναι ασύμβατα. Είναι συμπληρώ, συμπλήρωση στο το ένα στο κείμενο. Η έγκριση του πρώτου δεν αντιβαίνει σε οτιδήποτε από την επόμενη παράγραφο. Θα, θα είναι ε, β, και όχι γ, γ και όχι β, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Δεν είναι ασύμβατα. Ε, στο μικρόφωνο να μιλάτε πρόεδρε. Ο κύριος Γκουαλτιέρη ζητά να ελέγξουμε αν η τροπολογία 71 που θεωρώ ασύμβατη γιατί εγκρίθηκε το 70 είναι ενδεχομένως να έχει δίκιο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 δεν θυμάμαι που είχαμε φτάσει. Στο Y δεν είχαμε ψηφίσει την 72. Τέλο πάντων, τι να ψηφίσουμε για καλό και κακό. 72. Υπέρ κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Συμβιβαστική Y υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Που καλύπτει 76-77 Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 κατά πέπ, καταπίπτει το ίδιο το 80, 79 επίσης και το 81 άρα τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος να ψηφιστεί 81 Συγγνώμη. Πολύ καλό ο Γκουαλτιέρη, όλα τα θυμάται και τα καταλαβαίνει. Βλέπω το καντούκ καταπίπτει και μπερδεύομαι, αλλά η 81 δεν ψηφίζεται εάν είναι, αν εγκριθεί η 78. Ε, συγγνώμη, για ποια τροπολογία μιλάμε. Την 81, καλά λέω. Η 78 δεν ψηφίστηκε γιατί είχε καταπέσει. Άρα η γραμματεία δίνει τη νομική συμβουλή ότι ψηφίζουμε την 81 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέραση ψηφοφορίας. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ωραιότατα. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά υποχρεωτικά. Άρχεται ψηφοφορία. Βεβαίως ονομαστικά προφανώς. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Κάποιος που δεν θέλει να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 12 υπέρ, 4 κατά, 7 αποχές. Ωραία. Τελειώσαμε. Έχουμε για κάτι, με αυτό το θέμα έχουμε για κάτι ακόμα ψηφοφορίες. Πολύ σημαντική. Έκθεση Γκουαλτιέρη για το Μητρό Διαφάνειας που θα ψηφίσουμε. Συμβιβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει. Η τροπολογία 2. Β. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι πηγαίνουμε Στην τροπολογία 6, μαζί με την προφορική τροπολογία του εισηγητή, που εγώ ως συντάκτης τροπολογίας δέχτηκα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 7 καλύπτεται από τη συμβαστική. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω 10 υπέρ κατά απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 Βίλαντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 Σέπλιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 Hefner υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται εγκρίνεται εγκρίνεται αν θέλετε να κάνουμε την ε, ψηφοφορία για το 18 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας κρίνεται. Η 19 υπέρ κατά απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 περισσότερο πρέπει να είναι υπέρ του 21 κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα προχωρούμε στην 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Αλλά ας τσεκάρουμε λίγο το... την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπέρ. Ε, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40-41 καλύπτονται από τη συμβιβαστική C. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 καλύπτεται επίση από τη συμβαστική C. 44. Αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε. Μα εγώ το απέσυρα. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ όχι δεν ψηφίζουμε 49 γιατί καταπίπτει 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 μπορείτε να μας ψηφίσει, να ξαναψηφίσουμε. Γιατί ε, σηκωνόντουσαν και κατεβαίναν τα χέρια ταυτόχρονα, ε, πήγατε γρήγορα. Τη 45 σας παρακαλώ πολύ. Ας πω, ότι αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Ηλεκτρονικά. Για τη 45 λέμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο, ηλεκτρονικά, Πα, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το 90. Ψηφίζουμε την έκθεση Μπούζιτς. Λέγε να la relatrice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 Ah sì, sì, va bene, va bene. Sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora pongo in votazione. È stato ritirato. Bisogna chiedere a David Martin se... Risulta ritirato a me su questo. Λοιπόν, εδώ στο δικό μου χαρτί η τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. Συμφωνεί ο εισηγητής. Ορίστε. Λύθηκαν όλα. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4. Πέρας. Και εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 όχι έχει εγκριθεί το 2. Ψηφίζουμε όμως την τροπολογία 3 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την τροπολογία 6 γιατί ήταν ταυτόσιμη. Τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Θέλει κάποιος το λόγο? Τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια συνάδελφε Μάρτιν. Και νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε με τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι ήδη μεσημέρι. Πρόεδρος, παρακαλώ τους συναδέλφους, παρακαλώ τους συναδέλφους να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί έχουμε ε, την ε, συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Γιώζεφ Βάιλερ, ο οποίος είναι εξωτερικός προσκεκλημένος. Μη μας εγκαταλείπετε δηλαδή. Θα συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης.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 Allora riprendiamo i nostri Έχουμε καθυστερήσει αρκετά, ζητώ συγγνώμη και δημοσίω από τον ε, καθηγητή κύριο Βάιλερ, ο οποίο αναγκάστηκε να περιμένει εκτό ε, αιθούση. αλλά ξέρετε είχαμε ψηφοφορίε πάνω σε τρει εξαιρετικά σημαντικές εκθέσεις και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να διακόψουμε την, την ψηφοφορία αυτή. Ε, εδώ θα ξεκινήσει τώρα μια δημόσια ακρόαση, την οποία διακαώς επιθυμούσαμε, γιατί αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα ενδεχόμενα, τα σενάρια, τα οποία ε, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Θα συζητήσουμε ε, με, την, με βάση μια έκθεση που αφορά την, το μέλλον της Ευρώπης. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Ζόζεφ Βάιλερ, καθηγητή, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, τον οποίο γνωρίζουμε και από παλαιότερη ακρόαση. Ο κύριος Βάιλερ ξέρουμε ότι είναι αναφορά όσον αφορά ε, τέτοια θέματα. Υπήρξε ε, και ε, καθηγητή στην έδρα Ζαμονέ του Χάρβαρτ ε, και επίσης ε, καθηγητής σχολή, στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της ε, Νέας Υόρκης και μάλιστα ήταν σύμβουλος και στην Συνταγματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας, πρέπει να τελειώσουμε στη μία και μισή. Θα κάνουμε δύο συνεδρίες στην πρώτη συνεδρία θα δώσουμε το λόγο στον καθηγητή κύριο Γιώζεφ Βάιλερ να κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να αισθανθώ σαν όπως όταν μεταξύ των λεόντων ή αντίστροφα Έρχομαι όμως με κάθε ταπεινότητα και σεμνότητα ενώπιον σας ε, για να κάνω λόγο για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στους εκπροσώπους στο τέμενος της Δημοκρατίας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αναφέροντας ένα θέμα το οποίο αποτελεί φαν, φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 1979 με τις πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο ήταν η συμμετοχή μικρότερη από το 60%, μικρότερη από το μέσο όρο της συμμετοχής στις εκλογές στα κράτη-μέλη. Διαρωτήθηκαν γιατί δεν ε, υπήρξε κίνητρο να συμμετάσχουν περισσότερο οι Ευρωπαίοι τότε. Η απάντηση που δόθηκε ήταν «Μα γιατί να νοιαστούν να ψηφίσουν οι πολίτες αν και όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τόσο περιορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες». Και η πρόβλεψη ήταν ότι καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτούσε όλο και ευρύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες, τότε το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων θα αυξανόταν διότι αυτό ήταν εκείνο το οποίο ήταν το σημαντικό στοιχείο. Αν δεν είχε αρμοδιότητες δεν θα ενδιαφερόντουσαν οι πολίτες. Αν είχε θα ενδιαφερόντουσαν. Το θέμα το οποίο παρακολουθεί διαρκώς ως φάσμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι το γνωστό φαινόμενο ότι μεταξύ 1979 και 2009 οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εξουσίες του αυξήθηκαν δραματικά και δίκαια κιόλα. Και όμως ε, η ε, συμμετοχή στην, ε, στην επιτυχία των εκλογών μειώθηκε και στις τελευταίες εκλογές το 2009 ήταν περίπου το ίμιση εκείνων που συμμετείχαν από ποσοστό συμμετοχής το 1979. Να το πούμε ομά, όσο περισσότερες εξουσίες κέρδιζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο λιγότερο απέβαινε το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων. Υπήρξαν πολλές επεξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο. Κάποιες από τις πιο τυπικές είναι ότι πρέπει να επεξηγούμε τα πράγματα καλύτερα, λέει στους πολίτες. Δεν μου αρέσει αυτή η επεξήγηση. Έχει μια γεύση αρχαιομαρξισμού, παλαιομαρξισμού και σε σχέση με τον Μπρέχτ, αφού απογοητεύουν οι πολίτες του κυβερνώντες, σας αλλάξουν οι κυβερνώντες τους πολίτες. Έχει μια τέτοια συνοδευτική υπόγευση, μια εναλλακτική επεξήγηση θα έπρεπε να αναζητήσουμε για να δικαιολογηθεί αυτό το φαινόμενο. Στον πυρήνα, στην ίδια την καρδιά της δημοκρατίας βρίσκεται η επιλογή ως θεμελιώδες στοιχείο. Αν δούμε όλα τα δημοκρατικά στοιχεία, για παράδειγμα <clears throat> το γαλλικό προεδρικό σύστημα, το γερμανικό, το ιταλικό, το βρετανικό, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν όλες τις δημοκρατίες. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι δύσκολο να πιστούν οι πολίτες να εμπλακούν σε μια δημοκρατική διαδικασία και αφορούν επιλογές και τα δύο. Όταν πάνε να ψηφίσουν οι πολίτες τι γίνεται. Θεωρούν ότι κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ψηφίζουν αυτόν που θα τους ε, κυβερνήσει μελλοντικά. Και δεύτερον, επιλέγουν και ψηφίζουν σε κάποιο βαθμό πώς θα επιθυμούσαν να διακυβερνηθούν. Αν το μεταφράσουμε αυτό υπό πολιτικού όρους στην πολιτική επιστήμη, είναι η αρχή της λογοδοσίας και η αρχή της αντιπροσώπευσης αυτά τα δύο θέματα. Και τέθηκε το πρώτο αντίστροφο. Όταν πάει κανείς να ψηφίζει, τι γίνεται πρέπει να μπορεί να διώχνει τους ανίκανους και να μπορεί να αλλάζει την κυβέρνηση και τους κυβερνώντες και άλλοι να τους διαδέχονται ώστε να κυβερνήσουν τους πολίτες. Και θέλει κανείς να πιστεύει μέσα από όλα αυτά, αν αρκετοί πολίτες δηλαδή μπορέσουν να ψηφίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως εσύ ο πολίτης και να επιλέξει με αυτόν τον τρόπο, θα έχει αυτό επιπτώσεις στο πώς θα διακυβερνηθεί η χώρα και οι πολίτες. Αν υπάρχει μια κεντροαριστερή πλειοψηφία σε ένα κοινοβούλιο, ε, η πολιτεία θα ακολουθήσει μια κεντροαριστερή κατεύθυνση στις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Αν υπάρχει κέντρο, ε, δεξιά πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, ε, τότε οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν θα έχουν μια κεντροδεξιά κατεύθυνση. Αντιλαμβάνονται οι πολίτες τους συνασπισμούς ε, δεν πρόκειται για μια άμεση μετάφραση επιλογών σε πολιτικές, αλλά υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες των πολιτών. Ότι με την ψήφο μου μπορώ να αλλάξω τους κυβερνώντες, ε, αυτούς που με κυβερνούν. Μπορώ να διώξω, να αποπέμψω τους ανίκανους ε, και τους διεφθαρμένους. Και με, κάθε, με κάποιο τρόπο έτσι συμμετέχοντας και ψηφίζοντας στη δημοκρατική διαδικασία μπορώ να διαμορφώσω τα πράγματα όπως εν μέρει επιθυμώ εγώ. Πρόκειται λοιπόν για το ίδιο το DNA, το χαρακτηριστικό πυρήνα της δημοκρατικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στοιχείο σε σχέση με αυτό. Αυτά τα δύο λοιπόν θεμελιώδη ζωογόνα στοιχεία της δημοκρατίας δεν επικρατούν. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή στην πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι ψηφοφόροι πάνε, συμμετέχουν και αν ψηφίσουν με τον τρόπο που επιθυμούν μπορούν να διώξουν τους ανίκανους και τους διεφθαρμένους. Διότι δεν είναι δομημένη η Ευρώπη έτσι. Δεν είναι ένα κράτος. Παρότι ασκεί αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει πολλές φορές μια, ένα κλασικό κράτος, μια πολιτεία εντός εισαγωγικών. Και αν πάρουμε κάποιον σαν για παράδειγμα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σίγουρα δεν είναι ένας πρωθυπουργό, αλλά κάποιος που μπορεί να ασκήσει μεγάλη τα μάλα ε, επιρροή δεν υπήρχε διασύνδεση ή τουλάχιστον πολύ απόμακρη σύνδεση σε σχέση με τις ε, ε, ευρωεκλογέ για το ποιος θα πέρε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από διαβουλεύσεις του Συμβουλίου κατέληγε στο να επιλεγεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Η αρχή λοιπόν της αντιπροσώπευσης δεν ισχύει και δεν, δεν έχουν την αίσθηση οι πολίτες όταν ψηφίζουν ότι θα ψηφίσουν αυτός που θα, αυτόν που θα τους κυβερνήσει και θα αποπεμφθούν οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι λοιπόν σε σχέση με αυτές τις αρχές από μακρά μπορούν να εφαρμοστούν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ λίγοι με το χέρι στην καρδιά θα έλεγαν ότι υπάρχει η προοπτική σε σχέση με τις εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο ότι όταν κάποιος θα εκλεγόταν μέσω αυτών των εκλογών ως Ευρωβουλευτής θα ίσχυαν όλα αυτά. Και δεύτερον δεν υπάρχει καμιά επιστημονική μελέτη που να έχει αποδείξει ή καταδείξει μια συστηματική διασύνδεση μεταξύ μιας πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή της πολλαπλότητας, πολυμορφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε κέντρο αριστεράς είτε κέντρο δεξιάς και της πολιτικής κατεύθυνσης που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτίμηση των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές δεν μεταφράζονται συστηματικά και αυτόματα με αυτόν τον τρόπο στο επίπεδο της άσκησης πολιτικών και κατευθύνσεων πολιτικών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν αυτό αποδεδειγμένο απο, επιστημονικά. Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Μπορεί να, στη θεωρία να αναφέρεται κάτι τέτοιο, αλλά σε σχέση με μια κεντροδεξιά πλειοψηφία, για παράδειγμα στο Ευρωκοινοβούλιο, να έλεγε κανεί ότι, α, ορίστε, μια τέτοια πολιτική ασκήθηκε στην Ευρώπη, ε, μια και ήταν το Κοινοβούλιο, είχε αυτή τη διαμόρφωση. Και έχουν δίκιο οι πολίτε λοιπόν. Διότι όταν δεν αποκομίζουν το αίσθημα ότι ψηφίζουν και επηρεάζουν τα, ε, όσα τεκταίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο ή ψηφίζουν και επιλέγουν του κυβερνώντε του, ε, δεν μπορούν να πιστούν ότι ψηφίζουν και αποφασίζουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Ευρώπη. Γι' αυτό σε σχέση λοιπόν με τις ευρωεκλογές αποβαίνουν μια άλλη κρατη... ένα εγχείρημα ε, εκλογών σε ένα κράτος μέλος και έτσι εκφράζονται οι πολίτες. Αυτό ίσως θα μπορούσε να αλλάξει και θα άλλαζε με πολύ σημαντικό τρόπο με αυτά τα οποία κάνατε εσείς για αυτές τις πρόσφατες ευρωεκλογές, για αυτές τις ε, πρώτων θυρών ευρωεκλογές τώρα θα μπορούσαν να αλλάξουν διότι αυτά υπήρχαν ως ιδέα αλλά οι Ιταλοί έχουν μία παροιμία που λέει ε, νέα συζητούν, ένας όμως από αυτούς δραστηριοποιείται και πράττει κάτι. Οι πολλοί συζητούν ο ένας ε, δραστηριοποιείται. Και έτσι δόθηκε λοιπόν συνέχεια σε αυτό και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ακολούθησαν αυτή την κατεύθυνση. Το να πει κανεί τώρα ότι στι ευρωεκλογέ για το κοινοβούλιο, το επόμενο ευρωκοινοβούλιο, έμεσα θα είναι και μια προσφορά στου ε, πολίτε ε, για να ψηφίσουν τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ίδιοι με την ψήφο του. Ήταν ένα στίχημα αυτό. Ένα πρόταγμα που τέθηκε ως στίχημα δέχτηκαν οι πολιτικές ε, ομάδες, κάθε ομάδα είχε έναν υποψήφιο και στην προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει και θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα αμέσω. Δεν θα είναι μόνο μια εκλογή, δεν θα είναι μια εκλογή όπως παλαιότερα. Στους πολίτες ε, είπαμε ότι το κόμμα ή η ομάδα που θα κερδίσει τις εκλογές και εδώ υπάρχουν μικρά ερωτηματικά πως και ποιοι όταν κερδίσουν τις εκλογές τι θα κάνουν θα οδηγήσουν στην, ε, ακριβώς στην επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής στο μέλλον. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η πολιτική σημασία και εμβέλεια όλων αυτών και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχονται σε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα είναι ένα ορόσημο αυτό και είναι ένα ορόσημο διότι και είναι ενδιαφέρον αυτό που ε, διευθετήθηκε χωρίς αλλαγή της συνθήκης. Είναι η πιο σημαντική αλλαγή από οποιαδήποτε κίνηση προς τον εκδημοκρατισμό. Και αυτό ενδυνάμει αυτό που κάνει για την ευρωπαϊκή δημοκρατία συνεισφέρει περισσότερο από ότι οποιαδήποτε προηγούμενη πρωτοβουλία όπως το εγχείρημα για το Σύνταγμα της Ευρώπης που απέτυχε κατά το παρελθόν. Διότι εν δυνάμει δημιουργεί την δυνατότητα ε, προσφοράς επιλογής για τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους ώστε να επηρεάσουν τα πράγματα στον πυρήνα του δημοκρατικού ευρωπαϊκού συστήματος. Δεν υπάρχει λοιπόν δημοκρατία χωρίς αυτά τα στοιχεία. Με όλα τα πράγματα επικουρικότητα και όλα τα λοιπά, διαφάνεια, δεν είναι αυτά όλα η πραγματική επιλογή. Η δημοκρατική εμπλοκή και συμμετοχή και ο καθορισμός με αυτόν τον τρόπο είναι η επιλογή. Για πρώτη φορά θα υπάρξει η επιλογή αυτή, όχι για τον κυβερνώντα μας, διότι μπορούμε να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας ή ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως μια προσωπικότητα που έχει μεγάλη επιρροή στο αξίωμα που ασκεί. Και έτσι αυτό έχει τη σπουδαιότητά του. Πολλά μπορούν να πάνε στραβά βέβαια. Τι μπορεί πρώτα απ' όλα να πάει στραβά. Παράδειγμα, να είναι όπως τα καλυστία, ένα είδος διαγωνισμού καλυστίων διότι θα επιλέξουν μεταξύ υποψηφίων για την Προεδρία, αλλά όχι μεταξύ πολιτικών που θα τεθούν προς επιλογή. Πολλά εξαρτώνται από τα μέσα του τύπου. Ο κύριος Σούλτς και ο κύριος Γιούγκερ θα πρέπει επανειλημμένα να ερωτώνται στις συνεντεύξεις που δίνουν σε κάθε δημόσιο φόρουμ. Γιατί πώς ψηφίζοντας υπέρ ημών, κύριε, και όχι υπέρ του άλλου, του αντιπάλου σας, Πώς αυτό θα συνεισέφερε ώστε να δημιουργήσει τη διαφορά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Να τους υποχρεώσουμε δηλαδή να αρθρώσουν τον, τους λόγους για τις διαφορετικές πολιτικές ή διαφορετικές κατευθύνσεις που στοχεύουν να οδηγήσουν την Ευρώπη προς αυτήν. Όχι να πούν όχι, εγώ είμαι ένας ικανότατος πολιτικός που είναι και οι, και οι αντίπαλοι τους είναι, αλλά πώς ψηφίζοντας υπέρ ημών κύριε θα έκανε τη διαφορά για την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον σε σχέση με την υπερψήφιση του αντιπάλου σας. Αν δεν γίνει αυτό θα υπάρξει απογοήτευση. Απογοήτευση θα είναι ένα είδος καλυστίων που δεν θα δίνει καμιά νοηματικά δικαιολογημένη, ας το πω έτσι, ε, κινητοποίηση στους πολίτες υπέρ της μίας ή άλλης επιλογής. Δεύτερον, θα είναι υποχρεωμένοι να δεσμευθούν να δράσουν και να διαμορφώσουν την κατεύθυνση των πραγμάτων. Οι εξουσίες ε, και οι ε, αρμοδιότητες τους ως Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι περιορισμένες. Είναι συλλογικό σώμα το σώμα των Επιτρόπων. Θα μπορούν να τοποθετηθούν επί προγραμματικών διαφορών λοιπόν αν θα έχουν τη βούληση ασκώντας τις εξουσίες που έχουν υπό τη συνθήκη να διαμορφώσουν τις πολιτικές ως συλλογικού σώματος της Επιτροπής ώστε να υπάρχει μια πολυμορφία υπέρ της ε, κατεύθυνσης α ή β που θα έχουν επιλέξει γιατί διαφορετικά η υπόσχεση που θα έχει δοθεί ότι θα κινηθούμε προς αυτήν ή την άλλη κατεύθυνση δεν θα μπορεί να τηρηθεί. Είναι ένα νέο λοιπόν πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο και έτσι πρέπει να υποχρεωθούν να τοποθετηθούν. Και μετά θα υπάρχει και η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ίδια πολυμορφία, η ίδια πλειοψηφία για την εκλογή του Προέδρου σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Αν όλα αυτά σώρη και προϋποθέσεις ισχύσουν θα είναι πολύ διαφορετική η Ευρώπη που θα ακολουθήσει από την Ευρώπη που γνωρίζαμε. Διότι θα υπάρχει ένας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα έχει εκλεγεί με έμεση εντολή των Ευρωπαίων πολιτών τον ε, βασιζόμενο σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα τον διαφοροποιεί εκείνον ή εκείνην τον έναν ή τον άλλο από τους αντιπάλους με μια επιτροπή που θα έχει δεσμευτεί να κινητοποιήσει και να κινήσει την Ευρώπη προς την δεδομένη αυτή κατεύθυνση και μια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρόμοια θα δεσμεύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι στόχοι θα μπορούν να επιτευχθούν. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ελέγχων και αντι, αντιστάθμισης ε, και ε, πολλαπλής αντιστοίχησης. Ε, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να πάει στραβά, να μην δώσουν την προσοχή τους όπως θα έπρεπε οι πολίτες σε όλα αυτά. Είναι μια ξεχωριστή πολιτι... Ε, ένα ξεχωριστό ενδεχόμενο αυτό. Δεν ξέρω σε σχέση με το τι γίνεται σε σχέση με την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την, άλλη, τη μία ή άλλη χώρα. Πολλά εξαρτώνται από το είδο τη προεκλογική εκστρατεία, από τα μέσα του τύπου, την απήχηση όλων αυτών. Και δεύτερον, μπορεί να υπάρξει ω παρεμπίπτουσα επίπτωση να μην υπάρξει αύξηση τη συμμετοχή των πολιτών. Αν δεν υπάρξει αυτή η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, μειώνεται η νομιμοποίηση όλων αυτών και μειώνεται η κοινοβουλευτική διάσταση στην ε, επιρροή των πραγμάτων. Αν η συμμετοχή αυξηθεί και αυξηθεί ε, αισθητά και σημαντικά όχι κατά μία, δύο, τρεις ε, ε, ποσοστίες μονάδες αλλά επί κάποια, κάποια μεγαλύτερα ποσοστά τότε θα αυξηθεί αυτή η συνιστόσα. Μπορεί ένα κόμμα να μην κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Ε, λοιπόν ποιος θα είναι ο νικητής. Θα είναι αρκετά επιδέξιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ελιχθεί και να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα προς ε, την εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως θα έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί αυτή η συμμετοχή και επιρροή και όχι μόνο υπέρ του ενός ή άλλου ε, ε, υποψηφίου αλλά λόγω της ε, ψήφου των εχθρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς ευρωπαϊκών κομμάτων και θα υπάρξει μια πολύ πιο ζωντανή και κινητοποιημένη εκστρατεία για να μην ταπεινωθούν τα κόμματα αυτά σε σχέση με τα εχθρικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κόμματα σε σχέση με την εθνική, τον εθνικό συσχετισμό τους. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε ο εκλογικός κύκλος συμμετοχής να είναι μεγαλύτερος και αυτό θα σήμαινε μεγαλύτερη συμμετοχή, αν υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή τότε θα στεφτεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα βαθύτερο ερώτημα. Είναι έτοιμη η Ευρώπη για όλα αυτά, για μια πολιτικοποιημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι σήμερα τι συνέβαινε τα καλά ήθη, τα χρηστά ήθη όσον αφορά την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοσμοθεωρία της εκπροσωπούσε το σύνολο της Ευρώπης επρόκειτο για πολιτική μέσω κομματικής έκφρασης ε, χωρίς ιδεολογική όμως απόχρωση νομιμοποίηση απέρε από την επαγγελματική επιδεξιότητα και ικανότητα και τα αποτελέσματα των πολιτικών που επιτυγχάνονται. Όταν ε, επιλέγεται λοιπόν ένας πολιτικός ε, για να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεκδίεται των προηγούμενων κομματικών δεσμεύσεων, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι πλέον χριστιανοδημοκράτης, σοσιαλδημοκράτης, φιλελεύθερος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το ηθικό πλαίσιο που νομιμοποιούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι δεν ήταν ένα κομματικό σώμα ή πολιτικοποιημένο κόμμα, ε, πολιτικοποιημένο σώμα. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους ε, ε, κομματικές δεσμεύσεις. Δεν εκπροσωπούσαν ένα κόμμα, εκπροσωπούσαν μια χώρα, π.χ. τη Γερμανία. Δεν πεζόταν το παιχνίδι των κομματικών πολιτικών. Δεν γινόταν κάτι δεκτό. Το πείραμα στο οποίο λοιπόν απεκδίεται τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια σημαντική αλλαγή ως ορόσημο διότι αν στεφθεί με επιτυχία με τους τρόπους που προεξέθεσα και ακολουθήσει και το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται μέσω μιας εκλογής τύπου καλυστίων αλλά υπάρχει δέσμευση με ένα πρόγραμμα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με υποστήριξη του Συλλογικού Σώματος των Επιτρόπων και υποβοήθηση και στήριξη του Κοινοβουλίου αυτό θέτει το ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι και όριμοι για αυτή την πολιτική Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το αντίτιμο και το, το αντίτιμο για αυτή την Ευρώπη. Χωρίς να υπάρχει αυτή η κομματική δέσμευση. Αυτό θα σημαίνει μια τελείως διαφορετική Ευρώπη από αυτή που γνωρίζαμε και γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Οι παρεμβάσει ήταν σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Δίνω το λόγο τώρα στον καθηγητή κύριο Εμμανουηλίδη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών. Μας ανέφερε ο κύριο Εμμανουηλίδης ότι οι συνάδελφοί του, Φίσερ από το Ίδρυμα Μπέτεσμαντ και ε, από το Ίδρυμα Μποντουέν δεν είναι παρόντες. Μετά την παρέμβαση του κ. Ιβανοηλίδη θα παρουσιάσει, θα έχετε το λόγο και για τις δύο εκθέσεις. Ο κ. Μανουηλίδης έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και εσάς και την Επιτροπή σας που με κάλεσε να έρθω εδώ για να μιλήσω για πιθανές στρατηγικές επιλογές για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο, ακόμη περισσότερο ε, δηλώσει από τον καθηγητή κ. Βάιλε, αλλά θα προσπαθήσω να ξεπεράσω το πλαίσιο των ευρωεκλογών και να σας παρουσιάσω κάποιες πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον επόμενο πολιτικό κύκλο τα επόμενα έτη. Αυτό που συζητούμε είναι κομμάτι ενός ευρύτερου ε, πλαισίου που είναι ένα νέο, μια νέα σύμβαση για την Ευρώπη υποστηρίζεται από 11 ιδρύματα και προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε πιθανές εναλλακτικέ λύσεις, όχι σενάρια, για το πού θα είναι η Ευρώπη τα επόμενα 5-10 χρόνια. Εναλλακτικέ είναι, δεν είναι σενάρια και ε, τι συζητούμε με πολλού από εσά. Κάνουμε 40 με 50 εκδηλώσει, σε 16 γραφτά κράτη-μέλη. Ο κ. Σέφλιν ήταν σε μια τέτοια εκδήλωση στη Βουδαπέστη πριν λίγες εβδομάδες για να ακούσουμε τι απόψει και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, να παρουσιάσουμε ιδέε και συστάσει μαζί με μια ομάδα ατόμων που, έκαναν αυτές τις, που διαμόρφωσαν στρατηγικές Δύο πράγματα λοιπόν θέλω να κάνω το επόμενο διάστημα, να τι περιγράψω και να πω παραπέρα για να τις ενσωματώσω σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Για να δούμε πού προχωρούμε με την υφιστάμενη κατάσταση τώρα. Ποιες είναι οι πέντε εναλλακτικέ αυτές λύσεις. Να σας πω κάποιες σκέψεις μου πρώτα για το πού βρίσκεται κατά την άποψή μου η Ένωση αυτή τη στιγμή. Κατάσταση της Ένωσης. Σε αυτή τη φάση είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψουμε το πού βρισκόμαστε. Οι ιστορικοί στο μέλλον μάλλον θα μπορέσουν να αποτιμήσουν τι σημαίνει αυτή η τελευταία πενταετία, επταετία και η κρίση για την ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Δεν ε, είναι δεδομένο ότι οι σιδηροί νόμοι όπως αποκαλούν της Ευρωπαϊκής Ενωπής θα λειτουργήσουν εκ νέου, δηλαδή ότι θα προχωρήσει η Ένωση βάσει των πιέσεων, διότι η κρίση έχει μια σειρά παράπλευρων απολειών που θα παραμείνουν τα επόμενα έτη. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 12 προφανώς. Μετά την δράση και της Ευρωπαϊκής και Κεντρικής Τράπεζας και άλλων, συστημικά η κατάσταση φαίνεται καλύτερη Και λέω συστημικά γιατί αν πάτε για παράδειγμα στην Ελλάδα την ε, χώρα προέλευσής μου και πω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη τώρα θα μου πούν με δουλεύεις διότι η ανεργία των νέων είναι 60% το 1 τρίτο της, ε, του ΑΕΠ έχει χαθεί δεν μπορεί να πας να λες ότι η κατάσταση συστημικά είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά την επόμενη φάση της ενοποίησης, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα. Δεν είναι σαφές προ ποια κατεύθυνση θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα έτη και την επόμενη περίοδο. Και εδώ μπαίνουν οι πέντε στρατηγικές εναλλακτικέ λύσεις. Θα τις παρουσιάσω με κάπως αντικειμενικό τρόπο και στρατηγικά. Στο κείμενό μας υπάρχει πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πρώτη επιλογή είναι αυτό που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσω την, παραγω... Ε, παρομοίωση με το κυβότιο ταχυτήτων. Όπισθεν. Πίσω στα βασικά. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό που έγινε στο παρελθόν ήταν υπερβολικά φιλόδοξο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα γίνει δεν θα προχωρήσει σε μια στενότερη ένωση όπως λέει η συνθήκη και ούτε πρέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει οικονομική και πολιτική ένωση και θα έπρεπε να κάνει αναστροφή, να διδαχθεί από τα λάθη της, να επανεθνικοποιήσει ίσως κάποια στοιχεία, να διαλύσει την Ευρωζώνη από την παρούσα κατάσταση και εδώ και να σταθεί στο κέντρο της, ενιαίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ενιαία αγορά. Η προσδοκία δηλαδή δημιουργίας μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης δεν επιτευχθεί και θα οδηγήσει σε κατάρρευση. Άρα να μην κάνει μάταιες προσπάθειες να διορθώσει τα αδιόρθωτα, αλλά να ξαναγυρίσει του βασικού βασικούς της στόχους. Δεύτερη επιλογή. Νεκρό για να χρησιμοποιήσουμε το κυβότιο ταχυτήτων. Η Ένωση κινείται λόγω του παρελθόντος, των παρελθουσών δράσεων, μεγάλες προσπάθειες να δημιουργηθούν περιορισμένα, να δημιουργεί περιορισμένη τραπεζική ένωση, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ε, τώρα δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Τα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη, αυτοί που υποστηρίζουν την επιλογή αυτή λένε ότι τα κράτη-μέλη είναι αρνητικά, η κοινή γνώμη είναι αρνητική και το να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κατάσταση. Να μην αρχίσουμε να αναθεωρούμε τη συνθήκη, να σταθούμε σε αυτό που στην πολιτική επιστήμη λέμε νομιμοποίηση των νεκρών. Η τρίτη επιλογή είναι η ταχεία πορεία προς τα εμπρός. Μεγάλη ταχύτητα, αποδεχόμαστε ότι οι, τα επιτεύγματα του παρελθόντος δεν αρκούν, χρειάζεται περαιτέρω ενοποίηση και μέτρα για την εμβάθυνση της ένωσης της, της ενοποίησης της ΩΝΕΣ και ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στο κοινό καθώς και μια έντιμη συζήτηση, συζήτηση που δεν είχαμε τα τελευταία 3-4-5 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πολλές αποφάσεις λαμβάνονταν και κλεισμένο των θυρών. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προχωρήσουμε πιο φιλόδοξα, χωρίς να δημιουργήσουμε νέες διαιρετικές τομές, που σημαίνει ότι αν χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις συνθήκες, να αναμορφώσουμε το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Τούτο πρέπει να γίνει με συμμετοχή όλων των κρατών. Αυτό προφανώς απαιτεί συνένεση, συμβιβασμού, αλλά αποφεύγει νέες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πυρήνα και μη πυρήνα. Τέταρτη επιλογή. Τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Η ομοσπονδιακή προοπτική θα την πούν κάποιοι. Εμείς με επίγνωση δεν χρησιμοποιήσουμε τον όρο ομοσπονδιακό στην έκθεση. Μιλούμε για μια πλήρη οικονομική, πολιτική, δημοσιονομική και κοινωνική ένωση. Δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση με το όνομα κυβέρνηση, ένα νομοθετικό όργανο με ισχυρότερες εξουσίες για τη λήψη αυτόνομων αποφάσεων που εκφράζουν πραγματικά ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα. Μία ιδιότυπη ομοσπονδιακή ένωση και ξεπέρασμα της αντίφασης ενιαίου νομίσματος και εθνικών ε, συμφερόντων. Δημιουργία πολιτικών δομών που πάει παραπέρα και από ε, αυτό που περιέγραψε για τις συνέπειες της, ε, των επόμενων ευρωεκλογών καθηγητής κύριος Βάιλερ. Και αν δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη έτοιμα να προχωρήσουν μέχρι εκεί και υπάρχει μόνο μία, ένας πυρήνας που θέλει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή, να του επιτραπεί να προχωρήσει, έστω και αν αυτό σημαίνει να δημιουργηθεί μία ένωση του ευρώ, όπως ε, προτείνει η ομάδα Γκλίνεκε. Η πέμπτη εναλλακτική είναι αλλαγή της λογικής. Μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Εδώ ξεπερνιέται η παραδοσιακή συζήτηση, οι περισσότερες ή λιγότερες, λιγότερες Ευρώπης. Οι προηγούμενες εναλλακτικέ που προνέφερα είτε προς τα πίσω είτε προς τα μπρος, πηγαίνουν προς την λογική των, της πολιτικοποίησης, προσωποποίησης και κοινοβουλευτικοποίησης της Ένωσης. Η εναλλακτική αυτή λέει η προσέγγιση αυτή είναι απο, ε, απλουστευτική. Πρέπει να ξεπεράσουμε την ε, απλουστευτική λογική. Να φέρουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο το εθνικό πλαίσιο. Ακόμα και μετά από πολλά χρόνια δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό δήμο, έναν ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, μια ευρωπαϊκή λίγουα φράγκα και γιατί να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό δήμο όταν και οι εθνικοί δήμοι δεν λειτουργούν επαρκώς. Άρα πρέπει να προωθήσουμε νομιμοποίηση με μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινού, ε, με τοπικά δημοψηφίσματα, με θεμελιώδη δικαιώματα και μέτρα προστασίας. Αυτές είναι οι πέντε εναλλακτικέ. Επιστροφή, παγίωση, θαραλέα πρόοδος τεράστιο άλμα ή αλλαγή της ευρωπαϊκής λογικής. Στο τέλος, να σας δώσω και ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεν θα το βρείτε αυτό στην έκθεσή μας. Από μένα προέρχεται αυτό. Πού είμαστε. Και πάλι θα προσπαθήσω να σας πω τι προτιμώ, αλλά να δώσω μία ανάλυση θέτοντας την παρούσα κατάσταση στο πλαίσιο των εναλλακτικών που περιέγραψα. Το σαφές είναι ότι είναι σαφές προς τα που θα πάμε. Αλλά πηγαίνουμε μάλλον προς την ε, δεύτερη εναλλακτική. Στερεώνουμε, παγιώνουμε ό,τι έχουμε πετύχει. Κάποιοι λένε να γυρίσουμε πίσω για την επανεθνικοποίηση, αλλά δεν είναι πολύ. Η προώθηση προς ένα ποιοτικό άλμα δεν βρίσκει πλειοψηφία. Άρα η στερέωση των επιτευγμάτων είναι αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Μην το πάρετε λάθος, υπάρχει κίνηση. Το ότι υπάρχει ας πούμε συμφωνία για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης ή τη δημιουργία ε, αυτών που κάποιοι αποκαλούν ως συμβατικές συμφωνίες. Δείχνει ότι υπάρχει κίνηση, αλλά πέραν αυτών δεν γίνονται πολλά. Αν δείτε τι ζητάει η Επιτροπή στο σχέδιό της. Ή αν δείτε την έκθεση των τεσσάρων προέδρων υπό την ε, αιγίδα του κυρίου Φανρομπάη, πολλά από αυτά έχουν ήδη φύγει. Δεν μιλάμε για ένα ενιαίο πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων, για ένα ενιαίο πρόγραμμα ε, εγγύησης, ε, μια σειρά. Άρα, στην ουσία, πάμε στην δεύτερη εναλλακτική. Τα κράτη δεν θέλουν να πάνε παραπέρα γιατί φοβούνται ότι θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας μέσω μιας συνέλευσης ή μιας νέας συνθήκης. Υπάρχει ο φόβος του κόστους της συνένεσης. Τι σημαίνει να θέλεις να πετύχει συνένεση μεταξύ 28 κυβερνήσεων κρατών μελών για να αναθεωρήσει τη συνθήκη. Υπάρχει ο φόβος αποτυχιών στην επικύρωση. Υπάρχει το τραύμα του συντάγματος ε, που παραμένει και ο φόβο του τι θα γίνει αν υπάρξουν δημοψηφίσματα σε κάποια κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα ωστόσο τα κράτη θέλουν να κρατήσουν ε, να, να, να, να, λειτουργεί ο κινητήρα της μεταρρύθμιση, να κουνιέται το αυτοκίνητο. Και το βλέπουμε. Αν ακούσετε προσεκτικά την, ε, τι είπε η κυρία Μέρκελ που ανέφερε την ανάγκη αλλαγή τη συνθήκη, χωρί να μιλά όμω συγκεκριμένα για το περιεχόμενο ή τη διαδικασία της αλλαγής των συνθήκων ο κινητήρας της μεταρρύθμισης λειτουργεί αλλά στο ρελαντί. Γιατί θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό ήταν ο στόχος και του παρελθόντος. Να κερδίσουμε χρόνο για να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και το ερώτημα είναι, και εδώ τελειώνω, χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο. Υπάρχει ανάγκη να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος. Όταν, ξεκινήσα, όταν σταματήσαμε στη δεκαετία του 80 και του 90 ε, την πορεία προς το ενιαίο νόμισμα γιατί δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα και εγώ φοβάμαι, ε, θεωρώ ότι ο φόβος, ο βασικός φόβος είναι ο κατακαιρματισμός η υπόλωση θα την αποκαλέσουν κάποιοι κατακαιρματισμός μεταξύ ένωσης και πολιτών οικονομικός κατακαιρματισμός μεταξύ κρατών μελών, ετερογένεια, ολοένα και αυξανόμενη ετερογένεια μεταξύ των οικονομιών και έλλειψη εμπιστοσύνης, αύξηση της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και στο εσωτερικό των κοινωνιών. Κάτι που πριν λίγα χρόνια δεν φανταζόμουν ποτέ. Οι ερευνητές για τα εθνικά στερεότυπα ε, κατηγορούν ένα τον άλλον για αυτή την ε, μη προβλεφθήσα εξέλιξη και κατακαιρματισμός, διέρεση μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων. Κάτι που ενθαρρύνει την ό,τι πια δύναμη είναι αντί. Ίσως να χρειάζεται να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι από το να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τα κεκτημένα μόνο. Το ερώτημα, εσείς θα το συζητήσετε, γιατί όπως είπα στην αρχή, πάνω σε αυτό θα κάνουμε περαιτέρω δουλειά με συγκεκριμένε ιδέε. Γι' αυτό είμαι εδώ και περιμένω να έχουμε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους δύο καθηγητές και για την εισαγωγή που έκαναν. Έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτο ο κύριος Σαφλίνγκ. Παρακαλώ κύριο Σαφλίνγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο σας. Μου άρεσαν μου άρεσε η συγκέντρωση του καθηγητού Βάιλερ στις επιλογές της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό. Εγώ θα προχωρούσα ακόμα παραπέρα δέχομαι ότι υπάρχουν στοιχεία στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, που δεν ταυτίζονται με αυτά που ανέφερε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ε, ο κύριος Εμμανουλίδης και εγώ έχουμε συζητήσει τα πέντε σημεία τα οποία ανέφερε ήδη στη Βουδαπέστη. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι υπάρχει μία μείωση της νομιμοποίησης ε, της ευρωπαϊκής, της ενωσιακής ε, εξουσίας, πολιτικής δύναμης μάλλον. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, διάφορες εξτρεμιστικές και λαϊκίστικες δυνάμεις οι οποίες περιορίζουν τη δημοκρατία. Ωστόσο, αν υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες δεν ικανοποιούνται, τότε πραγματικά διανύουμε, διατρέχουμε μάλλον τον κίνδυνο πρόκλησης της δημοκρατίας. Πάνω απ' όλα, αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι υπάρχει ανερχόμενη ανισότητα ε, η οποία οδηγεί σε άδικη κατανομή της δικαιοσύνης. Και βεβαίως, ε, σωστά ή λάθος, ε, με το δάχτυλο δείχνεται η Ευρώπη σαν ένοχος. Τώρα, το θέμα της συμμετοχής στις εκλογές, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω εάν ξέρετε την εργασία του Ντόλα Σαββουά η άνοδος της κοινωνίας των πολιτών, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, όλων αυτών των ε, πολιτικός δρόντων κατά κάποιο τρόπο, ε, έχουν, χωρίς να είναι πολιτικοί, έχουν κατακαιρματίσει λίγο την πολιτική εξουσία. Και αυτό θα πρέπει να ξεπεραστεί ή τέλος πάντων να μελετηθεί ως πολλαπλασιαστικό φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ βέβαια θα συμφωνήσω και με την ανάλυση σας ότι όλοι ε, θέλουν να γίνει πιο νομιμοποιημένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό τουλάχιστον δεν έχει γίνει και ίσως μέχρι ένα βαθμό έγινε το αντίθετο. Το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να υποβάλω είναι ρητορικό βέβαια. Γιατί, γιατί υπάρχει αυτή η μία αναγνώριση της, ε, ε, του ευρωπαϊκού πολιτικού πεδίου η απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η δέσμευση. Εάν είσαι ας πούμε πολίτης ή ομάδα πολιτών ε, με πολιτική εξουσία σε, ευρωπαϊκό, ε, σε πολιτικό επίπεδο δεν, υπάρχει, δεν, δεν υπάρχουν έτσι, ευρωπαϊκά μονοπάτια τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε εύκολα. Κάνετε και μία πρόταση, δηλαδή ότι το μέγεθος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος ε, και με τον τρόπο αυτό ε, και αυτό το βρήκαμε, το είδαμε, ήταν έβριμα και της, ε, του, του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος ότι απομακρύνονται από την Ευρώπη και απομακρύνονται και από τις άλλες χώρες. Και αυτό το λέω και από τη δική μου εμπειρία στην Ουγγαρία. Τελευταίο σημείο. Επανέρχομαι μέσω αυτού στα όσα είπατε για την Κομισιόν που βλέπει τον εαυτό της σαν να είναι πάνω από την πολιτική. Αυτό είναι ανοησία βέβαια. Και βεβαίως είναι πολιτικό όργανο και η Κομισιόν και πρέπει να ορίσει τον εαυτό της σαν τέτοιο. Ε, αυτό που με ανησυχεί είναι αυτή η τάση που έχει μέρος της Κομισιόν να βλέπει τον εαυτό της πάνω από την πολιτική και πέρα από την πολιτική, ε, ενώ συζητάει με μία καθόλου εύληπτη τεχνοκρατική γλώσσα. Το τελευταίο σημείο, ήταν το πρώτο τελευταίο αυτό που είπα τώρα, αφορά την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, ε, ένα θεσμικό πλαίσιο προ-παγκοσμιοποιημένο δεν έχει λάβει υπόψη τον πολλοπλασιαστικό ρόλο όλων των πολιτικών ε, ε, πρωταγωνιστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που με απασχολεί τώρα είναι η βιωσιμότητα της ήπιας δύναμης, soft power σε αυτόν τον παγκοσμιωμένο κόσμο. Βλέπουμε ας πούμε και με την περίπτωση του Πούτιν πώς ε, αντικρούεται η ήπια δύναμη. Η ήπια δύναμη μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γκουελτιέρη είχε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Ξεκινώντας με τον κύριο Εμμανουηλίδη, θα έλεγα ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική επιλογή που επικρατεί είναι η δεύτερη πολιτική επιλογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. για τις ε, διεργασίες που προηγήθηκαν με τις αποτυχίες που συνδέονται σε σχέση με την ε, ε, Δημοσιονομική Ένωση όσον αφορά αυτούς τους πυλώνες ως άξονες σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων που διαγράφονται κάποια θέματα από την διαβούλευση και στο τέλος δεν απομένουν πολλά. Και ακόμα και όταν διαρωτόμαστε για το τι έγινε και τι κάνουμε με την Τραπεζική Ένωση με το SRM αν ολοκληρωθούν και στεφθούν με επιτυχία που θα είναι μείζον ε, και κτημένο αυτό. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι είναι ένας περίπλοκος σύνθετος μηχανισμός πολιτικών όρων και προϋποθέσεων που δημιουργούν την, το συμπέρασμα ότι επικρατεί δεύτερη επιλογή Είχαμε και εκπρόσωπο της ε, Βρετανικής κυβέρνησης ε, και για τη θέση της μη διεξαγωγής ε, δημοψηφίσματος από πλευράς των εργατικών για κάποια συμφωνία ισορρόπησης των πραγμάτων μία λογική των πραγμάτων από τους μεν και τους δε αυτή η λογική δεν είναι όμως από ό,τι φαίνεται η πιο ρεαλιστική Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να πω αν διαφοροποιήσουμε την επικρατούσα πολιτική επιλογή ως ε, προτίμηση αυτή που υιοθετείται από τους πολιτικούς ηγέτες και προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στις διαργασίες και διαδικασίες ε, πέρα από την συνειδητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτικά εμπλεκόμενων θα έλεγα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ε, αισιόδοξοι για το ε, εναλλακτικό σενάριο το οποίο οδηγεί στην αλλαγή και μεταβολή ήδη τώρα αυτών των ε, εναλλακτικών λύσεων. Αφενός ε, αληθεύεται αυτό το οποίο αναφέρθηκε ως πολιτική πρωτοβουλία από πλευράς του κυρίου Βάιλερ διαδραματίζει ένα ρόλο αλλά και για την εσωτερική δυναμική των πραγμάτων των μηχανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Παράδειγμα, αναφορά στο θέμα ότι και αυτό υποστήριξε η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων για να υπάρχει ένας υποψήφιος από πλευράς ε, των κομμάτων για αυτό το αξίωμα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση χωρίς αλλαγή της συνθήκης. Πρέπει να δει όμως και τα πράγματα προηγούμενα σε σχέση με τα όσα ίσιαν. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας φυσικά χωρίς την πολιτική βούληση, πολιτική πρωτοβουλία ε, και σε σχέση με τα όσα είχαν ε, συμφωνηθεί προηγούμενα μπορεί αυτό να μην είχε υιοθετηθεί και σε σχέση με τη διατύπωση του άρθρου 77 υποβοηθήθηκαν τα πράγματα προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν, υποβάλλει, δεν επιβάλλει κάποιον ε, ε, υποψήφιο. Υπάρχουν τα αποτελέσματα των εκλογών που πρέπει να λαγγλυφθούν υπόψη με τις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν περαιτέρω. Βρέθηκε λοιπόν και μια βάση με βάση τη συνθήκη ένα άρθρο και με την πολιτικοποίηση των πραγμάτων που ίσως μελλοντικό ιστορικός θα μπορούσε να σταθμίσει και να κρίνει. Ε, έχουν ξεκινήσει ίσως κάποια πράγματα και νωρίτερα σε σχέση με όλα αυτά όσα είπατε στην παρουσίασή σας εν μέρη, χωρίς δηλαδή πλήρη συνειδητοποίηση των πολιτών, όλα αυτά συνέβησαν κατά την κοινοβουλευτική αυτή θητεία. Είχαμε μια σαφή κεντροδεξιά πλειοψηφία, πλειοψηφία και ένα σαφή προσανατολισμό σε σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πάλι καθιστά πιο ενδυναμωμένη την πρόταση να πει κανείς ότι αν τώρα υποστηρίξουμε και κάνω λόγο φυσικά ως ε, ε, σοσιαλιστής αν υποστηρίξετε εμάς τους σοσιαλδημοκράτες και τον Σούλτς ως υποψήφιο θα υπάρξει μια αλλαγή διότι αυτό το οποίο μετρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την σταθερότητα, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης φυσικά δεν ήταν μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πράγματα τα οποία κινήθηκαν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και όλων ημών και με εκλογέ και την ε, κεντροδεξιά πλειοψηφία σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Τώρα αλλάζει η στάθμιση των πραγμάτων, η ισορροπία των πραγμάτων με βάση τις φημομετρήσεις και μετά όσα συμβαίνουν σε σχέση με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Σημαντικές αλλαγές, σημαντικά κεφάλαια της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε όλη αυτή τη διεργασία συνολικά αυτή η ιδέα των υποψηφίων είναι μια πολιτική πρωτοβουλία αλλά είναι και κάτι το οποίο ερμηνεύει μια προσέγγιση που είχε ξεκινήσει ήδη κατά το παρελθόν δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται απόλυτα με τα τρία π που προανέφερε ο κύριος Εμμανουηλίδης στην ε, εισαγωγή του. Αλλά το θεσμικό πλαίσιο μέσα στη θεσμική δυναμική των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα βαθύτερο ρεύμα πραγμάτων από ό,τι συνειδητοποιεί κανείς με μια πρώτη ματιά και σε σχέση και με τους πολιτικούς ηγέτες. Η κυρία Μέρκελ η ίδια κάποιους μήνες πιο πριν είχε πει ποτέ δεν θα δεχθούμε μια τέτοια λύση των υποψηφίων ε, που ε, θα εκπροσωπούν τους πολίτες όσον αφορά το αξίωμα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δυναμική λοιπόν αποδείχθηκε στεναρότερη και ισχυρότερη από ό,τι πίστευαν κάποιοι. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και στο γεγονός στη συνέχεια ότι υπό τους όρους περιεχομένου ουσίας της μεταρρύθμισης και με την λογική της παγίωσης, ε, εμπέδωσης αυτών των πραγμάτων ίσως μπορέσουμε να υπερβούμε με μια ισχυρότερη προώθηση προς τα εμπρός και ένα, μια, ένα βήμα προόδου να αλλάξουν πολλά πράγματα με την διαδικασία πολιτικοποίησης, κοινοβουλευτικοποίησης της εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεισφέρει αυτό το βήμα στη μεταβολή και αλλαγή του πλαισίου λογικής των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να αλλάξει και τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά τις επιλογές σε σχέση με τα κρατούντα κατά το παρελθόν και ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό. Ο κύριος καθηγητής Βάιλερ επεσήμανε πολλά προβλήματα πρακτικού χαρακτήρα θέματα και ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν θα έρθει η χρονική στιγμή υλοποίησης και εφαρμογής όλων αυτών που προαναφέρθηκαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο γίνεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 θα διοργανώσει ένα δείπνο και μετά οι πολιτικές ομάδες θα διοργανώσουν ένα πολιτικό, ας το πω ε, πλαίσιο κατά την επομένη πρωία. Ακόμα και αν αυτό το πλαίσιο Δηλαδή μπορεί να αναγνωστεί ως η βούληση να μην χάσει την πρωτοβουλία και το πάνω χέρι το Συμβούλιο, ο αποφασιστικός παράγοντας ε, μετά τις εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Η διασύνδεση δηλαδή των ευρωεκλογών με την απόφαση, λήψη απόφασης σε ένα πλαίσιο δέσμης μέτρων ως πακέτου. Δηλαδή η απόφαση για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πακέτο θα πρέπει να ρυθμιστεί με τον πρόεδρο του, ε, ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του αξιώματο του κυρίου Φαν και του αξιώματο της υπά του εκπροσώπου, του υπά του εκπροσώπου που έχει αυτή τη στιγμή η κυρία Άστον, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα των εκλογών σε αυτή την εσωτερική θεσμική ισορροπία και με έναν αναλογικό μηχανισμό εκπροσώπησης ανάλογα με τα πόσα μέλη θα έχει κάθε ομάδα μεταξύ της ε, Κιανής ε, και ε, Ερυθράς στήλη μετά τις εκλογές αυτό θα έχει την επιρροή του άμεσα σε σχέση με την επιλογή αυτών των αξιωμάτων. Αυτό θα αποτελέσει ίσως και ένα μεθεπόμενο κίνητρο για τις ε, ε, ακόλουθες με, ε, μεθεπόμενες ευρωεκλογές περαιτέρω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία μεταρρύθμισης και αναθεώρησης και συνταγματικά, στη συνταγματική συνιστόσα των τεκτενόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταβάλουν και να αλλάξουν και την ε, λογική των πέντε αυτών προτύπων που μας παρουσιάσατε στην εισήγησή σας. Ευχαριστώ. κύριος έχει το λόγο. Ο καθηγητή Βάιλερ είπε ότι σε όλε τι δημοκρατίε οι ψηφοφόροι έχουν δύο επιλογέ. Οι ψηφοφόροι έχουν δύο επιλογέ. Ποιο και πώ κυβερνώνται. Η... Το να μετατρέψουμε. Υπάρχει ωστόσο και το δεχόμενο κατά πώ οι ψηφοφόροι θα μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να ψηφίσουν τις, ε, να κυβερνώνται από τους ε, υπό, από τις ε, διάφορες εξουσίες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η αύξηση της, των εξουσιών του Κοινοβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύονται από μικρότερη συμμετοχή σε εκλογές. Μας είπατε ότι οι εκλογές του 2014 θα δώσουν στους ψηφοφόρους ε, τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων υποψηφίων για την Προεδρία της Επιτροπής. Η ιδέα αυτή είχε προταθεί από τον καθηγητή κύριο Μαντούρο πριν από δύο χρόνια εδώ. Στηριζόταν στην ιδέα ότι θα υπήρχαν εγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει εκλογικό σώμα της Ευρώπης με συλλογική ταυτότητα. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος. Υπάρχει βεβαίως ευρωπαϊκή πολιτιστική ή αρχαίγονη ταυτότητα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η προπαρασκευαστική δουλειά δεν έχει γίνει. Αυτό δεν είναι ιδεολογικό, αυτή η παρατηρήση δεν είναι ιδεολογική. Το ίδιο θα έλεγα και υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης να ήμουνα. Για παράδειγμα, Ρώτησα κάποιου ε, συνταξιούχου καθηγητέ πρόσφατα τι ήξεραν για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και με κοίταξαν κάπως χαμένοι. Κατόπιν του ρώτησα τι ήξεραν ως προς το ότι το Μάιο θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων υποψηφίων για τη θέση του Πρόεδρου τη Επιτροπή. Ακόμα πιο χαμένα με κοίταξαν. Δεν ήξεραν τίποτα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Βεβαίω, ήξεραν τι ήταν η Επιτροπή, και ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Μπορώ να σας πω ωστόσο ότι υπάρχει πολλοί κόσμος, στη Βρετανία τουλάχιστον, που δεν γνωρίζει την απάντηση σε καμία από τις δύο ερωτήσεις. Η κόρη μου έχει και μια μικρή ιστορία. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τη ρωτούσε ο κόσμος φίλη της τι κάνει ο πατέρας σου και έλεγε ότι είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του έλεγαν τι είναι τούτο. Αυτό μπορεί να είναι ευθύνη των μέσων στη Βρετανία. Δεν ξέρω. Το αφήνω κατά μέρο. Συνοψίζω. Μπορούμε να μεταφράσουμε τις ε, ψήφους, τις ευρωεκλογέ σε ψήφους για έναν υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής που θεωρείται ότι έλαβε αν όχι την πλειοψηφία ή αν μη τι άλλο την ε, σχετική πλειοψηφία αγνοώντας βεβαίως την ψήφο εκείνων που ψήφισαν εθνικά κόμματα και όχι ευρωπαϊκά κόμματα. Ωστόσο, θα είναι μια ψήφος που δεν θα ξέρουν ότι ψήφισαν οι ψηφοφόροι. Μια ψηφοφορία στα σκοτεινά χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει ε, το ψηφοδέλτιο θυμάστε όταν ε, έπαθε εγκεφαλικό ο αντιπρόεδρος κ. Παπαστάμκος, είχε πει ο κ. Σούλτς, ο κόσμος δεν ξέρει καν τι ψηφίζει. Αυτό τηρουμένου των αναλογιών μπορώ να σας το πω και για τις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ κ. Νταφ. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι με εκπλήσει σε σχέση με το μικρό μας αυτό πείραμα με, τους ε, υποψήφιους, τον, ανώ, τους ανώτερους υποψήφιους για αυτό το αξίωμα σε σχέση με μια ιδέα την οποία έχουμε συζητήσει επί 15 ετία. Δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η προσέγγιση προτού υπάρξει μια πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια με διεθνικούς, διεθνείς ε, ε, ε πίνακες υποψηφίων, καταλόγους υποψηφίων. Είναι όμως αυτό ένα ενδιάμεσο σημαντικό βήμα. Σημαντικό γιατί, διότι δημιουργεί και προέρχεται από το φεντεραλιστική προσέγγιση, ομοσπονδιακή προσέγγιση. Και αυτό σε σχέση όχι μόνο με τον Μάρτιν Σούλτς που επελέγει από πλευράς των σοσιαλδημοκρατών από έναν στενότερο, μικρότερο κατάλογο υποψηφίων αλλά επίσης και σε σχέση με τον Μισελ Μπαρνιέ που ήταν υποψήφιος για το ΕΛΚΑ και που ήταν θελκτικός και ένας, ε, έκανε μια ε, θελκτική εκστρατεία για να μπορέσει εκείνο να είναι ο υποψήφιος όμως ιτήθηκε από τον Ζαν ε, Κλόντιο Juncker και σε σχέση με μια ιστορική υποσημείωση πραγματικά θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς τις ικανότητες και τη θέση του κυρίου Μπαρνιέ. Όλα, όσα όλοι όσοι συμμετέχουν βρίσκονται υπό τεράστια πίεση διότι υπάρχει μετάθεση από την, ε, τους συμβιβασμούς μιας πολιτικής κοινοβουλευτικής ε, ε, ζωής στην δραστηριοποίηση ενός προεδρικού ας το πω έτσι πλαισίου και πώς τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία, θα βγουν από αυτή τη διαδικασία σίγουρα με το αντίτιμο το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν πληττόμενα θα οριμάσουν οπωσδήποτε. Και έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος καθηγητής Βάιλερ ότι το κλειδί θα είναι ο νέος αυτός πρόεδρος επιλέγοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει εκείνη την νομιμοποίηση πέρα αυτού εκείνη που δεν ίσχυε στο παρελθόν θα μπορέσει στη θέση αυτή που θα εκλεγεί να διαμορφώσει το συλλογικό σώμα των επιτρόπων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να ακολουθηθούν οι δικές του προτιμήσεις και κατευθύνσεις. Και είναι σημαντικό όχι επειδή είναι θέμα κομματικό αυτό, αλλά επειδή θα συμβολοποιήσει την ε, ουσιώδη ε, ένταση που θα οδηγήσει σε μια αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που θα επιθυμούσαν μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφενός και των άλλων που θα ήθελαν να ε, επικεντρώνονται τα πράγματα στο ε, Συμβούλιο. Αυτό το ζήτημα θα είναι το κέριο ζήτημα αντιπαράθεσης ε, κατά την επόμενη σύμβαση συντακτική συνέλευση που θα πρέπει να το εξετάσει και να το αναλύσει ως στοιχείο εκείνοι που θα ήθελαν να δουν τι θα μπορούσε να συμβεί με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μετατρεπόταν σε μια κυβέρνηση θα μπορούν τουλάχιστον <clears throat> να δουν την εφαρμογή της, των επιπτώσεων των όσων προτάθηκαν από πλευράς της ομάδας Πινέλη και της ομάδας Μπέρτεσμαν κατά το παρελθόν. Μια τρίτη παρατήρηση, παρατήρηση που έκανα καθώς ε, ε, έχω ρημάσει πλέον σε αυτό το επάγγελμα. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά στην αξιολόγηση και εκτίμηση των δημοκρατικών θεμάτων σε σχέση με τα κράτη-μέλη και μεταξύ κρατών μελών πολύ μεγαλύτερη και με περισσότερη διαφοροποίηση από ό,τι φαντάζονται οι πολίτες και υπό το πλαίσιο της εκλογικής νομοθεσίας και το πλαίσιο του πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι περιφέρειες και πώς θα πρέπει να γίνεται η χρήση δημοψηφίσματος ή δημοψηφισμάτων, δηλαδή στο συνταγματικό πλαίσιο και συνταγματική νομοθεσία και πρακτικές εφαρμογές όλων αυτών. Η πολυμορφία και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών είναι πολύ μεγάλοι και μεγάλες. Αλλά ταυτόχρονα δεδομένης αυτής της μεγάλης ε, ποικιλομορφίας ε, όπως αυτή εκτίθεται όλο και μεγαλύτερη ήταν η αίσθηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει και υφίσταται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους συνταγματικούς όρους του παιχνιδιού και τους πολιτικούς όρους των τεκτενωμένων για παράδειγμα για την ε, ανάμιξη σε θέματα που κατά το παρελθόν θα ε, θεωρούν εσωτερικές υποθέσεις ε, ενός κράτος μέλους και σε σχέση με τον κύριο Ρέντζι για παράδειγμα και την εκλογική νομοθεσία όπως ε, διαμορφώθηκε, διαμορφώνεται και προτείνεται και αν υπάρχει, υπάρχουν κάποιες επικρίσεις ε, που ε, έχουν γίνει και ασκηθεί από τους οπαδούς τους σε σχέση με την, τα όσα εγώ είπα από την Ιταλία και αυτό είναι τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης των πραγμάτων και υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική των πραγμάτων, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύουν οι πολίτες πολλές φορές. Το συμπέρασμά μου σε αυτή τη φάση της ε, εκλογικής εκστρατείας ε, είναι το εξής. Η πιο σημαντική μεμονωμένη απόφαση που θα πρέπει να λάβει το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι η εξής θα επιμείνουμε και θα εμείνουμε στην σύγκληση μιας συντακτικής συνέλευσης νέου. Σίγουρα θα υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή των συνθήκων. Αρκετές κιόλας ίσως κατά την περίοδο της επόμενης κοινοβουλευτικής εντολής και θητείας. Όμως η χρονική στιγμή και συγκυρία κατά την οποία η πλειοψηφία οι πλειοψηφίες και ο σύνθετος και πολύπλοκος χαρακτήρας και το θάρρος που θα απαιτείται θα είναι η λιδία λίθος που θα λειτουργήσει σε σχέση με την ψήφιση και την τοποθέτησή μας για την διεκδίκηση δικαιωμάτων από πλευράς μας μέσω μιας συντακτικής συνέλευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσω αυτού του εγχειρήματο θα πρέπει να δούμε τα συνταγματικά ζητήματα και προκλήσεις ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και έτσι θα πρέπει να πορευθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους συμφωνίας για την περίοδο, την εποχή μετά την επικράτηση των εθνικών ε, πολιτικών ε, σε ένα ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο και φυσικά σε σχέση με την προσπάθεια αυτή που έγινε, φεντεραλιστικού χαρακτηρισμού που έγινε, εν μέρει ήταν επιτυχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο σε άλλους τρεις συναδέλφους, αλλά θα, πρέπει να αφήσουμε και χρόνο στους, δύο καθηγητές ε, να ε, απαντήσουν, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε στη μια Πρέπει να αφήσουμε την αίθουσα και να ελευθερώσουμε και τους διερμηνείς ο συναδέλφος Μέλκοβιτς. Μπλάνκοβιτς. Μπλάνκοβιτς. Έλεγα και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βάιλερ και κύριε Εμμανουηλίδη. Ε, μας ε, ε δώσατε πολλά διαφωτιστικά σχόλια αναρωτιέστε ποια είναι η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2014. Η ανάλυση μου από πλευρά βέβαια κάποιου που προσπαθεί να, ε, που προσπαθούσε για 20 χρόνια περίπου να προσεγγίσει, να φέρει τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, η εξή. Πρόκειται για μια ρεαλιστική κατάσταση η οποία ε, φέρνει και τα τραύματα των πολλαπλών κρίσεων των τελευταίων 10 χωρών και την προσπάθεια πολλών χωρών να βρουν την ανεξαρτησία τους αλλά και μια τάση επανεθνικοποίησης των κρατών μαζί με είναι δημοκρατική νομιμοποίηση ε, των θεσμών και του πολιτικού κόσμου. Όταν ε, συζητάσαμε με πολίτες και τους μιλάς για ε, επανασυμφιλίωση και ανάπτυξη και τα λοιπά, πολύ συχνά τελικά σε ρωτάνε, ναι, αλλά ποια είναι η προστιθέμενη αξία για μένα. Όλο και περισσότερα ε, ας πούμε μπορεί να, η απάντηση να είναι ε, φέρνει κάποια θετικά στοιχεία σε οικονομικά και, και κοινωνικά ε, κριτήρια, σε οικονομικούς και κοινωνικούς όρους η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε από μία περίοδο που κανείς ε, δεν το ανέφερε βέβαια και εδώ θα μιλήσω σαν και μέλος της ε, Επιτροπής Προπολογισμών όπου κανείς ε, δεν ανέφερε τρία πράγματα. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε μία σε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο χαμηλότερο σε νούμερα και ποσά από τις προηγούμενες φορές. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και δεν είναι δυνατόν να το αποφύγουμε. Δεύτερον, όσον αφορά τη διεύρυνση. Η Κροατία κατάφερε ε, να μπει και είναι η πρώτη χώρα μετά την Ελλάδα, λέει ο ομιλητής. Και τα μέλη, οι χώρες οι οποίες είναι κοντά στη δικιά μου, είναι η Σλοβενία, είναι η Ουγγαρία, είναι η Σλοβακία, είναι τώρα η Κροατία και ίσως μία από τις παλιότερες χώρες ε, που πηγαίνει προς, τη, προς τις μελλοντικές ενδεχομένως χώρες. Ο τρίτος ε, φόβος είναι ο φόβος ε, των δημοψηφισμάτων. Δεν είναι μονάχα το θέμα της Νίκαιας και της Ελισσαβόνας για την Ιρλανδία. Το 2005 στη Γαλλία και στις κάτω χώρες που ακόμα έτσι ε, στοιχιώνει όλες τις συζητήσεις και όλο τον κόσμο. Δεν τα θέλουμε αυτά τα δημοψηφίσματα. Τα φοβόμαστε και κατά αυτή την έννοια η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών κομμάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα μάλιστα ε, εμείς ε, υπερψηφίσαμε τη δημιουργία και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων, πολιτικών κομμάτων είναι αυτή η προσπάθεια ε, να προχωρήσουμε προς μια καινούρια αρχή και είναι καλό βήμα αυτή η ε, εκλογή του Προέδρου της ε, Κομισιόν. Και όπως υπόθηκε και προηγουμένως, η Κομισιόν, πέρα και ξέχωρα από αυτό που λένε πολύ συχνά οι επικεφαλίστες της, είναι πολιτικό όργανο, κάνει πολιτική δουλειά και εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, κινητοποιηθούν ε, και ε, τα κυρίαρχα κατά κάποιο τρόπο πολιτικά κόμματα έτσι ώστε να αντιστρέψουν τις παρούσες τάσεις. Νομίζω ότι αυτά τα mainstream πολιτικά κόμματα της Ευρώπης πρέπει να μιλήσουν πλέον και νομίζω ότι ε, και ελπίζω μάλλον ότι η πρόβλεψη του καθηγητού Βάιλερ ότι τελικά η συμμετοχή στις ευρωεκλογές θα είναι μεγαλύτερη ελπίζω να ε, επαληθευτεί και αν ε, η πρόβλεψή σας είναι σωστή, τότε νομίζω ότι και η έκβαση για τα κλασικά πολιτικά κόμματα θα είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έφνερ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βάιλερ και τον κύριο Εμμανουηλίδη για τις πολύ επικοδομητικές και ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις τους ε, στις εισηγήσεις τους. Πραγματικά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για οτιδήποτε επετεύχθη και μπορέσαμε να επιτύχουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ταυτόχρονα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το εγχείρημα πραγματικά διακυβεύεται, τίθεται εν κινδύνο και εν αμφιβόλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η επιλογή υπαριθμών 2 μεταξύ των 5 που μας εκθέσατε είναι η πιο πιθανή να επικρατήσει. Ταυτόχρονα όμως θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να οπισθοδρομήσουμε ή να υπαναχωρήσουμε, αλλά τέλος δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω χωρίς να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προηγούμενο ώστε να ενταχθούν περισσότερο οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες στην Ευρώπη έχουν αποκομίσει την Ευρώπη <clears throat> ότι η Ευρώπη δεν είναι δική τους, δεν είναι οι ίδιοι, δεν τους, αντιπροσωπ... δεν τους εκπροσωπεί και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε τη σχέση δεσμού μεταξύ των πολιτών και της Ευρώπης. Να πούν ναι είμαστε η Ευρώπη εμείς, μπορούμε να συνεισφέρουμε να αλλάξει το πρόσωπο της Ευρώπης και αυτά είναι τα βήματα τα οποία ε, έχουν γίνει για παράδειγμα σε σχέση με τα πολιτικά πολιτικά κόμματα που ζητήθηκε να υποβάλουν προγράμματα και πλατφόρμες με υποψηφίους, με ανώτατους υποψήφιους Spitzenkandidaten ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τις, τους πολίτες ε, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν να μπορέσουν οι πολίτες να αισθάνονται ότι εκλέγουν τον ανώτερο υποψήφιο που επέλεξαν ώστε ο δικός τους ανώτερος υποψήφιος να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα. Κατανοώ την ιδέα πίσω ε, από την ε, ιδέα μιας μη πολιτικής ή πολιτικοποιημένης Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και όλο και λιγότερο είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να είναι και να γίνεται όλο και περισσότερο πολιτικό αυτό το πλαίσιο και να κινηθούμε, κινητοποιηθούμε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε με τις συνθήκες μεταξύ των ε, κρατών μελών και των ε, κρατών μας, ε, των αποφάσεων του Συμβουλίου και του διακυβερνητικού πλαισίου σε μια Ένωση που όλο και περισσότερο οι πολίτες θα έχουν την αίσθηση που θα αποκομίζουν ότι μάλιστα εμείς είμαστε εκείνοι που αποφασίζουμε προς τα που θα κινηθούμε και που θα πάμε. Όλο και περισσότερο λοιπόν αρμοδιότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο που στο τέλος, τέλος θα πρέπει να είναι στα χέρια των πολιτών να αποφασίζουν είτε άμεσα είτε μέσω της εκλογής στο Ευρωκοινοβούλιο των εκπροσώπων τους. Όλο και περισσότερο πρέπει να αποκλίνουμε από την διακυβερνητική συνιστόσα και προσπάθεια προσέγγισης των πραγμάτων σε μια δημοκρατικώς λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπέρ και χάρη των πολιτών. Και θα έλεγα ότι το να σταματήσουμε και να μείνουν στάσιμα τα πράγματα δεν είναι μια επιλογή για μας. Αυτό θα σήμαινε ότι θα χάναμε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από τους πολίτες μας και καθημερινά. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να ε, επιλέξουμε φιλόδοξα εγχειρήματα και προγράμματα <clears throat> να μην θεωρούν οι πολίτες ότι ε, εσείς είσαστε οι πολιτικοί, εμείς είμαστε οι θέατες. Όχι, οι πολίτες να συμμετέχουν έχουν την εντύπωση ότι διαμορφώνουν συμμετέχοντας τα πράγματα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα αναλάβει τα, το αξίωμά της, όταν θα υπάρξει το χρονικό, η χρονική ευκαιρία το 2015 να συγκαλέσουμε μια συνταγματική συνέλευση, να ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Και θα προσέθετα εκείνοι για παράδειγμα που φοβούνται ότι οι Βρετανικές προτάσεις ε, να ε, επιστρέψουν αρμοδιότητες και εξουσίες στα κράτη-μέλη ε, ή σε άλλα πεδία δεν θα πρέπει να μας κάνει να ε, διστάζουμε να εξετάσουμε τέτοια θέματα. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να εξεταστούν στη συνταγματική συνέλευση και με την πίεση ε, ενδεχομένως δημοψηφισμάτων ή των της διαβούλευσης μεταξύ μιας κυβέρνησης και μιας άλλης είναι σημαντικό να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Και είναι σημαντικό να συζητηθούν τα θέματα επιστροφής αρμοδιοτήτων και εξουσιών στα κράτη-μέλη ή σε ένα τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ακόμα και για αυτά τα σημαντικά θέματα χρειαζόμαστε περισσότερες αρμοδιότητες από την άλλη πλευρά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν αμφωτέρωθεν. Η ιδέα της σύγκλησης μιας ε, συνταγματικής συνέλευσης ε, και το άρθρο 48 της συνθήκης της Λισαβόνας είναι πολύ σημαντικές υποθέσεις. Πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα θετικά διαφορετικά από τις ε, προηγούμενες συνταγματικές συνελεύσεις. Ε, αυτό θα σημαίνει ότι χρειάζονται και περισσότερο, χρειάζεται και περισσότερος χρόνος για τη συνταγματική συνέλευση. Είναι δεδομένες οι δυσκολίες και δυσχέρειες για να συγκλίνουν οι παραδόσεις και οι διάφορες διαφορετικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να είναι θέμα ενός έτους ε, μόνο για παράδειγμα, αλλά ετών πολιετές εγχείρημα ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ώστε να δημιουργηθεί η νομιμοποίηση να θεμητοποιηθεί η συζήτηση και εξέταση αυτών των θεμάτων σε διαβουλεύσεις ε, λιγότερη χρονική πίεση που θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και με, όσον αφορά και τους κανονισμούς και διατάξεις για τη συντακτική συνέλευση σφάλμα ήταν το ότι δεν μπορούσε δημοκρατικά να ψηφίσει η συνταγματική συνέλευση αλλά ήταν η προεδρία της συνταγματικής συνέλευσης που θα αποφάσιζε για την τελική έκβαση των τεκτενόμενων και των πραγμάτων στη συνταγματική συνέλευση. Καλύτερη εμπλοκή και περισσότερη εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και αυτό ήταν τροτό σημείο της προηγούμενης συνταγματικής συνέλευσης. Και αν ένας συγκεκριμένος αριθμός πολιτών 400.000, 500.000 προσυπογράψουν ένα αίτημα όσον αφορά ότι θα ζητούσαν το ένα ή άλλο θέμα να το εξετάσει η συνταγματική συνέλευση θα έπρεπε αυτό να εξεταστεί από αυτήν. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνω. Η τελική επιλογή μέσω της ψήφου θα πρέπει να δοθεί στους πολίτες με την εμπλοκή τους. Θα γίνουν τέτοια δημοψηφίσματα. Π.χ. η Ιρλανδία, ε, Μεγάλο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Καλό θα ήταν να υπήρχε ένα δημοψήφισμα που θα διαμορφωνόταν όπου το Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελούσαν μέρος αυτού αλλά θα βρισκόταν υπό ευρωπαϊκούς κανόνες και κανονισμούς όταν θα διεξαγόταν και θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή συνένεση για μια πιο δημοκρατική και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν μια εφικτή πρόταση, μια μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι οι συνομιλητές μας δεν ενέταξαν τις σκέψεις τους για την Ευρώπη στο διεθνές πλαίσιο. Δεν μπορεί να δούμε πώς θα είναι η Ευρώπη και πώς θα χτιστεί χωρίς να την συσχετίσουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Η έκθεση για την ε, Ευρωαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, για παράδειγμα, είναι σημαντικό στοιχείο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μορφή ε, σχέση θα έχει η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, η τέταρτη εναλλακτική μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Έχω μία ερώτηση ωστόσο. Όταν συναντιόμαστε, τους, συναντάμε τους συμπολίτες, τους ψηφοφόρους μας, μας λένε τις τράπεζες τις σώσατε, εμάς όχι. Η εναλλακτική τέσσερα πώς θα αντιμετωπίσει το την κοινωνική διάσταση. Ποια κοινωνική Ευρώπη είναι δυνατή. Επίσης, μιλάτε για την χρήση κάποιου, για την ε, συνεργασία κάποιων κρατών μόνο για να προχωρήσουν. Υπάρχει η ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό είναι ένα εργαλείο εφικτό. Τελευταίο θέμα. Η απογοήτευση των πολιτών συνδέεται με την ε, έλλειψη ικανότητας να καταλάβουν την Ευρώπη πολλοί πολίτες νομίζουν ότι η Ευρώπη είναι εξαιρετικά περίπλοκη, ένα μηχάνημα, ένας μηχανισμός που έχουμε δημιουργήσει και που δεν τον καταλαβαίνουν. Άρα γίνεται ζήτημα δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών που με εντυπωσίασαν στην ε, εμπειρία μου είναι ο αριθμό των μη νομοθετικών εκθέσεων. Μας πνίγουν οι νομο, μη νομοθετικές εκθέσεις, που σημαίνει ότι οι νομοθετικές εκθέσεις είναι λιγότερο ευανάγνωστες και επίσης πώς μπορούμε να ξαναδώσουμε την εξουσία, να δώσουμε την εξουσία πρωτοβου, νομοθετικής στο Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει παρέμβαση του νέου πρόεδρου της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Δίνω αμέσως το λόγο, γιατί πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, στον καθηγητή κύριο Βάιλερ. Πέντε λεπτά με τον έναν, πέντε με τον άλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Βάιλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να τα ακούω να ακούσω όλες αυτές τις αντιδράσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες. Να κάνω μία παρατήρηση ωστόσο. Έχω την εντύπωση πως το Κοινοβούλιο δεν εκτιμά ιδιαίτερα τις συνέπειες του τι έγινε με τους υποψήφιους ε, για την Προεδρία της Επιτροπής. Να το πω πιο δραματικά. Αν αποτύχει, δηλαδή, αν δεν κινητοποιηθεί κοινή γνώμη, αν δεν αυξηθεί η συμμετοχή, αν η συζήτηση δεν γίνει για πολιτικές και όχι απλά εθνικότητα, σε εθνικό, σε εθνικό επίπεδο, αν το Συμβούλιο δεν ακολουθεί την άποψη του Συνοβουλίου, το Κοινοβούλιο θα βγει σαφώς αποδυναμωμένο από τις ευρωεκλογέ. Η ικανότητά του να μιλήσει, να μιλά στην Επιτροπή και το Συμβούλιο θα είναι ακόμα πιο αδύναμη τότε από ό,τι σήμερα. Η ικανότητά του να λειτουργήσει ως η φωνή του λαού θα αποδυναμωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν το δοκιμάσαμε δεν δουλεύει θα αποδυναμωθεί το Κοινοβούλιο. Και όσο και να σέβομαι την κοινωνία των πολιτών και όλους τους άλλους, το κέντρο της δημοκρατίας είναι το Κοινοβούλιο πάντα. Ένα αποδυναμωμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αν πετύχει, αν το Κοινοβούλιο καταφέρει να κινητοποιήσει στην προεκλογική εκστρατεία και στις επιλογές, ιδίως δε στη συνέχεια που θα δοθεί ούτως ώστε δηλαδή να υπάρξει ένας πρόεδρος επιτροπής με πρόγραμμα, με επιτρόπους που θα υποστηρίζουν τις θέσεις του, με μια σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που θα ανατρέψει, που θα ανακατέψει την Ευρώπη βάσει των υποσχέσεων που θα έχουν δοθεί στο, ε, εκλογικό σώμα, θα είναι οι επιλογές 3, 4, 5 μαζί. Θα είναι μεγαλύτερη αλλαγή από τις διάφορες συνθήκες. Θα είναι μια πιο μεγάλη συνταγματική αλλαγή στην Ευρώπη από την εισαγωγή της ε, ε, ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Αποδυναμώνεται η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Είτε αποτύχει είτε πετύχει. Αν αποτύχει αποδυναμώνει το Κοινοβούλιο, αν πετύχει θα έχουμε μια τελείως διαφορετική Ευρώπη. Ο κ. Εμμανουηλίδης. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις παρατηρήσεις στα σχόλιά σας που ήταν ιδιαίτερα σκόπιμα και φυσικά δεν μπορώ όλα να τα καλύψω. Θα προσπαθήσω με τις σημειώσεις μου να κάνω τα εξή να επικεντρωθώ σε τρία πράγματα σχετικά σύντομα. Με τον ανώτερο υποψήφιο Spitzenkandidat ως θέμα. Θα έλεγα μάλιστα υπάρχει μεγάλη σπουδαιότητα και αυτό ευθυγραμμίζεται στο να υπάρχουν τέτοιοι υποψήφοι για αυτό το ανώτατο αξίωμα αλλά ταυτόχρονα να μην το υπερτονίζουμε να μην υπερτονίζουμε αυτή τη σπουδαιότητά του είναι ένα πείραμα, πείραμα όλο αυτό ένα πείραμα το 2014 σχετικά. Θα συναθούν συμπεράσματα και θα δούμε για το 2019 τι θα γίνει. Ένα σύστημα ίσως ε, υποψηφίων σε κάποιο κατάλογο. Τα πράγματα βρίσκονται διαρκώ υπό εξέλιξη, ενρευστό. Ναι, υπάρχει λοιπόν ευκαιρία πραγμάτων όπως είπε ο κύριος Βάιλερ και κάποιοι καν, κίνδυνοι αλλά και κάποια συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να συναχθούν μετά τις εκλογές για την Ευρωβουλή τον Μάιο και μετά την 25η Μαΐου, μετά τις τι θα γίνει με τη νέα Ευρωβουλή, πώ θα ξεκινήσουν αυτά τα πράγματα υποσυζήτηση σε σχέση με τα θέματα τα θεσμικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα πρέπει συνειδητά να λάβει μια απόφαση μέχρι πού θα φτάσει σε σχέση με τις επιπτώσεις αυτού του εγχειρήματο το Ευρωκοινοβούλιο έναντι των άλλων. Ανάλογα με την απόφαση που θα υιοθετήσετε ως Ευρωβουλή, τι επιπτώσει θα επηρεάσει αυτό το ευρωκοινοβουλιο εναντι των αλλων αναλογα με την αποφαση που θα υιοθετησετε ω ευρωβουλη αυτο θα επηρεασει αυτο το εγχειρημα με, τον, με τους υποψήφιους για το αξίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα μπορέσουν αυτές οι δυνατότητες να ευδοκιμήσουν στο μέλλον. Αυτό δεν είναι μια εξάπαντος προσπάθεια και τέρμα, τελεία και παύλα. Είμαστε σε μια ενρευστό ε, κατάσταση, με μετεξέλιξη πραγμάτων. Η ισορροπία, η συνταγματική των πραγμάτων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις και αξιολογήσεις για τα τελευταία 4-5 χρόνια, που ήταν μια έκτακτη συγκυρία, μια ξεχωριστή περίοδος κρίσης, που ουσιαστικά το εκτελεστικό υπέστη της ε, επιπτώσεις και οι εθνικές κυβερνήσεις και τώρα τι θα γίνει στο μέλλον και τι, πώς, αυτά θα απορρεύσουν ε, πρέπει να δούμε και σε σχέση με την συνθήκη της Λισαβόνας η, οποία συνέπεσε με την ε, κρίση αυτή θα, δεν θα πρέπει να βιαστούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα σε σχέση την παγίωση, εμπέδωση πραγμάτων ή μετακίνηση, κίνηση προς τα εμπρός. Εγώ, εμένα μου φαίνεται ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο ακινητοποιηθεί και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να μην μείνουμε ακινητοποιημένοι κινητοποιημένοι και να είμαστε πιο φιλόδοξοι κινητοποιούμενοι. Αυτό θα είναι θέμα και στρατηγικών επιλογών για πολλά κράτη-μέλη. Συνοψίζω, είναι δυσχερέ το εγχείρημα. Θα υπάρξουν διαφορετικέ αντιδράσει σε διαφορετικέ ε, χώρε. Τι χρειάζεται. Μέρος τη επιλογή ένα. λιγότερο οι Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο να επηρεάζουν και ακαθορίζουν τα πάντα. Χρειάζεται πρόοδος το να ακινητοποιηθούμε και να μείνουμε στάσιμοι δεν είναι επιλογή. Παρότι ο βαθμός, πόσο βαθιά είναι η κρίση και πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις, είναι πολύ μεγάλης διάστασης σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει η εντύπωση ότι είναι μεγάλη η κρίση και τα προβλήματα. Σε άλλα πιστεύουν ότι είναι μικρότερη η διάσταση αυτή από ό,τι κατά το παρελθόν. Η πίεση έχει ε, μειωθεί σίγουρα, όμως το να μείνουμε κινητοποιημένοι δεν είναι ε, επιλογή σωστή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί μια μεγάλη συναλλαγή, μια μεγάλη συμφωνία, deal, pact, συμφωνία, συνθήκη η δημιουργία ενός συμβιβασμού στο ανώτατο εφικτό επίπεδο, όχι στο χαμηλότερο. Το θέμα και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να φτάσει κανείς εκεί σε αυτό το σημείο. Ποια είναι η καλύτερη τακτική προσέγγιση για να το πετύχει. Λέγεται χρειάζεται μια συντακτική συνέλευση για να κινητοποιηθούν τα πράγματα, για τη δημόσια συζήτηση και διαβούλευση όλων αυτών. Αλλά υπάρχει μεγάλος, υπάρχουν πολλοί φόβοι να γίνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν λοιπόν, να ληφθούν απόλυτα υπόψη και να τα συνειδητοποιήσουμε πλήρως

σε σχέση με την μεταρρυθμιστική ε, ε, συνιστόσα των πραγμάτων ή προπαρασκευαστική φάση των πραγμάτων σε σχέση με το τι θα γίνει για τη συνταγματική συνέλευση και τις φοβίες που υπάρχουν. Επίτευξη κάποιων μεταρρυθμίσεων. Αλλά χρειάζεται και η ανάγκη να προετοιμαστεί, να προπαρασκευαστεί αυτή η συντακτική συνέλευση σε διαφορετικά επίπεδα. Να επιτευχθούν όμως και να προχωρήσουμε στην επίτευξη αρκετών ε, όρων και προϋποθέσεων για να πάψει να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη φοβία που υπάρχει υπάρχει ε, εν ώψη αυτού του, ε, αυτής της προοπτικής και σε σχέση με την Γερμανία για παράδειγμα, για το ποιες είναι οι επιθυμίες πραγματικά του, του Βερολίνου, υπάρχουν διαφορετικά μηνύματα και τοποθετήσεις. Υπάρχει όμως και η βούληση μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με τη μορφή και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζουν προς τα που θα κινηθούν και θα κινητοποιηθούν, αλλά υπάρχει η ανάγκη να γίνει αυτό. Τώρα, σε σχέση με τις ε, τα ερωτήματα που τέθηκαν προσωπικά θα έλεγα ο ρόλος της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, διαφορετικών ταχυτήτων. Πρέπει να το δει κανείς υπό λειτουργικότητα, υπό την πτυχή της λειτουργικότητας. Έχουμε ήδη μια διαφοροποιημένη, διαφορετική προσέγγιση μεταξύ αυτών των θεμάτων στην Ευρώπη, διαφορετική διαστρωμάτωση. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο, αλλά να είμαστε συνετοί και προσεκτικοί. Και όσον αφορά την ολοκλήρωση, διαφοροποιημένη ε, ολοκλήρωση, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτον είναι δύσκολο για μένα να καθορίσω ποιοι θα ήταν στον πυρήνα και ποιοι θα ήταν εκτός πυρήνα. Θα ήταν οι χώρες της Ευρωζώνης στον πυρήνα και οι άλλες εκτός. Για αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να σημειωθεί η πρόοδος αλλά να είμαστε προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε νέες διαχωριστικές γραμμές πράγμα το οποίο θα ήταν επιβλαβές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λίγα δευτερόλεπτα μας απομένουν μένουν για να σας ευχαριστήσω. Σας λέω ε, ε, ένα εγκάρδιο ευχαριστώ και να σας πω ότι είστε καλεσμένοι με τους αντιπροέδρους και τους συντονιστές ε, σε γεύμα στο εστιατόριο των βουλευτών. Ελπίζω να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ.